Good morning everybody. We have a long... Καλημέρα σα, κυρίε και κύριοι. Έχουμε μια μεγάλη μέρα. Παρακαλώ καθίστε και μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μα. Θα συνεχίσω λοιπόν στα γερμανικά. Ich will dich anfangen, hab's nicht. Αρχίζουμε την πρώτη ψηφοφορία εναρμόνιση της εσωτερικής αγοράς. Θέλετε να λάβετε το λόγο. Σύντομα παρακαλώ. Σύντομη θα είμαι. Αγαπητοί συναδελφοί, Θέλω να ευχαριστήσω για την καλή συνεργασία στα πλαίσια της γνωμοδότησης. Πολύ καλή και επικοδομητική συνεργασία είχαμε. Και η πολιτιστική διάσταση αναδείχθηκε όπως έπρεπε και ε, το παρατηρητήριο δεν θα παρακολουθεί μόνο τις απομιμήσεις και την πειρατεία, αλλά θα λαμβάνει υπόψη και πολιτιστικά θέματα. Ευχαριστούμε Ζαμπίνε. Έχετε το... Έχετε κείμενο με καλή σήμανση και σημειώσεις για να με παρακολουθείτε έτσι με γκρι χρώμα υπογραμμισμένα κλπ. Συμβιβαστική 1. Υπέρ. Όχι αυτή, όχι αυτή, την άλλη. Okay. υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 62 υπέρ κατά αποχές έλεγχος άρχεται ψηφοφορία επί της 62 πέρας 9 προς 15 απορρίπτεται. 63 έχει αποσυρθεί. 64 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 20 υπέρ, 5 κατά. Ε, συγγνώμη, άμα δεν φαίνεται καλά το χέρι σας πρέπει να κάνουμε έλεγχο. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά χέσα απορρίπτεται. Πάμε στην 66 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 71 υπέρ κατά αποχές Δεκτή. Από ήρθε 69. 72 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 73 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 78 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 79 υπέρ κατά αποχές δεκτή 80 υπέρ κατά αποχές έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία επί της 80 πέρας 15 προς 12 δεκτή 81 υπέρ κατά αποχές δεκτή 8 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 82 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 83 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 84 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 85 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 86 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 87 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 88 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 91 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 93 υπέρ κατά αποχές δεκτή 94 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται προφορική τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή 95 υπέρ κατά αποχές δεκτή 96 υπέρ κατά Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την 96. Πέρας. Απορρίπτεται 14 προς 14. 11 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 98 υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος. Την 98 άρχεται η ψηφοφορία. <coughs> Πέρας. 16 προς 12. Απορρίπτεται. 99 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 100 υπέρ. Κατά. Αποχές έλεγχος. Την 100. Ε, Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 15 προς 13. Εντάξει. Δεκτή. 101 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 102 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 105 υπέρ κατά αποχές έλεγχος την 105 ε, άρχεται πέρας 15 προς 13 υπέρ 106 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 109 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 110 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή. όχι τη 12, αφού δεχτήκαμε την 110. Ψηφίσαμε τζάμπα. 111 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 116 Μπαντή Κούτζετ υπέρ κατά αποχές δεκτή. 117 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 118 υπέρ κατά αποχές δεκτή 119 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 120 υπέρ κατά κατά αποχές απορρίπτεται 121 υπέρ κατά αποχές δεκτή 122 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία στην 122. Πέρας. 16 προς 12 δεκτή. 124 υπέρ. Κατά. Αποχές έλεγχος. 124. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 14 προς 13. 126 υπέρ κατά αποχές δεκτή 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή 17 Α, συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 23 υπέρ κατά αποχές δεκτή 24 υπέρ κατά Πάμε στην 25. Ναι, 25 ψηφίζουμε υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 26 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 27 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 29 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 30 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή 34 υπέρ κατά αποχές δεκ... απορρίπτεται 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 40 όχι, ε, όχι 37 υπέρ κατά αποχές δεκτή 38 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 40 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 39 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 41 υπέρ. Κα... 41 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 42 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία, δεύτερο τμήμα της 42. Πέρας. 17 προς 12 απορρίπτεται. 43 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 44 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβι... Όχι, την 45 θα ψηφίσουμε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 54 τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή, τελική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 22 υπέρ, 5 κατά, 2 αποχές. Ε, συγχαρητήρια Ζαμπίνε και συγχαρητήρια στους Σκιώδης. Προχωρούμε στο σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης, οι επιτρεπόμενες χρήσεις ορφανών έργων. Θέλεις να πεις κάτι παρόμοιο με το προηγούμενο Ζαμπίνε. Όχι, δεν θέλω να πω το ίδιο. Θέλω να πω ότι παρόλο που πήραμε τις δύο εβδομάδες, θέλαμε κι άλλο χρόνο για να επεξεργαστούμε με την προσοχή που άξιζε το θέμα αυτό. Και θα ήθελα ε, θα ήθελα κάτι ευρύτερο, να μην εστιαστούμε μόνο στα βιβλία και στα έντυπα, στην έντυπη βιβλιογραφία. Λυπάμαι γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό που την πολιτιστική μας βιομηχανία την επηρεάζει σε βάθος. Θα ήθελα περισσότερο χρόνο και νομίζω ότι εκφράζω όλους τους εισαγητές. Ευχαριστώ παρόλα τα αυτά όλους που κατέθεσαν τροπολογίες επικοδομητικές που συνεργάστηκαν με τόσο καλό τρόπο και στα πλαίσια του δυνατού πραγματικά προσπαθήσαμε να διευρύνουμε κάνουμε την οδηγία για να την κάνουμε πρακτική στην εφαρμογή και ελπίζω να ληφθούν υπόψη όσα θεωρούμε πολιτιστικά σημαντικά. Ευχαριστώ πολύ. Μη με κακίσετε για το θέμα του χρόνου. Η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή έθεσε κάποια όρια. Επίσης και η Κομισιόν έχει θέσει κάποια ε, όρια. Ίσως στο μέλλον θα έπρεπε να το λάβει υπόψη της η Κομισιόν αυτό και να δώσει περισσότερο χρόνο να προβλέψει γιατί θέλουμε να εργαζόμεθα ε, διεξοδικά σε βάθος και όχι επιλεκτικά. Και πραγματικά στη νέα εποχή τα βιβλία θα πρέπει να ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη. Ε, βλέπω ότι χαμογελάτε με πολύ φιλικό τρόπο. Λάβετε τα υπόψη όλα αυτά. Πάμε στην ψηφοφορία για τα ορφανά. Συμβιβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές ε, ξανά. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 134 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 138 υπέρ. Κατά αποχές ξανά. 138 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 139 υπέρ. Κατά. Αποχές έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 14 προς 16 απορρίπτεται. 140 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 141 υπέρ. Όχι, την 146 παρακάτω. 146 ναι, ναι, ναι. Ε, του, υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Ελέγχουμε την 146. Μπαρναράμπα του. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα στις ψηφοφορίες. 17 προς 14. Δεκτή. 148. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 147, 147 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 150. Έχει αποσυρθεί. 151. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 20. Την 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 152 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 153 υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία την 153. Πέρας. 22 κατά, 9 υπέρ, απορρίπτεται. 155 υπέρ, κατά. Ξανά. 155 υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 21 υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 154 υπέρ, κατά. Αποχές, έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία την 154. Πέρας. 14 προς 14 απορρίπτεται. 156 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 157 υπέρ. Ε, όχι, όχι, σε ένα τμήμα. 157 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 158 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 159 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 17 προς 14 εγκρίνεται. 160 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές Έλεγχος στο δεύτερο τμήμα του ε, της 160. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 27 προς 4 απορρίπτεται. 161. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές, έλεγχος, ελέγχουμε την 22 άρχητη ψηφοφορία. Πέρας. 20 υπέρ 10 κατά εγκρίνεται 166 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 168 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 176 να ελέγξω. Την 168. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Ψηφίζουμε την 168. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 15 προς 15 απορρίπτεται. 176 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Την 176 άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. 16 προς 14 δεκτή. 220 ε, ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Την 220. Πέρας. 17 προς 14 δεκτή. Προφορική τροπολογία 1 τώρα. 175 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 23 έχει αποσυρθεί. 177 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 24 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία την 24. Πέρας. 17 προς 10. Να σηκώνετε καλύτερα το χέρι. Κάνει και καλή γυμναστική. Δεκτή λοιπόν. Ή 25 υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 13 προς 18 απορρίπτεται. 26 ε, υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Πάμε στην άλλη σελίδα. 183 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 187 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 188 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 16 προς 15 δεκτή. 190 υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 23 προς 8. Δεκτή. Ε, συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τώρα πάμε στην άλλη σελίδα, στην 192. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 193. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 194 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 195 υπέρ κατά αποχές δεκτή 220 υπέρ κατά αποχές δεκτή πάμε τώρα στην τροπολογία 30 υπέρ κατά αποχές δεκτή 31 υπέρ κατά αποχές δεκτή πάμε στην άλλη σελίδα όχι, 32 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Την 32 ελέγχουμε. 32. Ψηφίζουμε την 32. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. 23 προς 7 δεκτή. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 34 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 35 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 36 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 37 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 219. 219 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 220 υπέρ κατά αποχές έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία στη 220. Πέρας. 18 προς 11 απορριπτεται ε, Πέμπτο τμήμα της 220 υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. 222 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 224 υπέρ κατά αποχές δεκτό 225 υπέρ κατά αποχές έλεγχος τη 225 άρχεται η ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας 17 προς 9 δεκτή Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Την τροπολογία 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 18 προς 12. Δεκτή. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 20 προς 10 δεκτή. 38 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 39 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 3 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 41 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 42 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 40 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Πάμε τώρα στην 47 που είναι κάτω. Ψηφίζουμε τη 47 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή 57 υπέρ Α, την 60 θα ψηφίσουμε υπέρ κατά αποχές δεκτή 61 υπέρ κατά αποχές έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία την 61 ψηφίζουμε πέρας 16 προς 15 απορρίπτεται 6 υπέρ κατά ξανά υπέρ κατά αποχές δεκτή 64 υπέρ κατά αποχές δεκτή 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή το κάτω υπέρ κατά αποχές δεκτή 9 υπέρ κατά αποχές, έλεγχος, την 9, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 17 προς 13 δεκτή. 73 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος Την 73. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 21 προς 10 απορρίπτεται. 74. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 77. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 78. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 82. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Προχωρούμε 89 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 100 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Την 100 ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. 14 προς 15 απορρίπτεται. 101 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 102 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 103 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 104 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Πάμε τώρα στη συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 114 υπέρ κατά αποχές έλεγχος στην 114. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 21 προς 10 απορρίπτεται, 115 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, συμβιβαστική 9 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 122 υπέρ, κατά αποχές έλεγχος, άρχεται η ψηφοφορία, την 122 ψηφίζουμε, πέρας της ψηφοφορίας, 15 προς 16 απορρίπτεται, 123 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 227 υπέρ κατά αποχές έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία πέρας 19 προς 12 δεκτή 228 υπέρ κατά αποχές έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία πέρας 16 προς 15 δεκτή 229 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 230 υπέρ, κατά, αποχές έλεγχος, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 21 προς 10 απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 27 ψήφοι υπέρ, κανείς κατά τέσσερις αποχές, θερμά συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Ωραία. Θυμίζω, 11 και 4 έχουμε την Επίτροπο. Ησυχία παρακαλώ. Ησυχία παρακαλώ. Συνάδελφοι, στις 11 και 4 θα έρθει η Επίτροπος. Παρόλα αυτά θα ήθελα να πω ότι έχετε λάβει πρόσκληση για συζήτηση με τους βραβευθέντες με το λογοτεχνικό βραβείο την επόμενη εβδομάδα. Οπωσδήποτε θα είναι ενδιαφέρον ε, στην ε, βιβλιοθήκη να συζητήσετε με τους συγγραφείς αυτούς. Επίσης ε, θυμίζω ένα εξαιρετικό έργο για το Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ. Χθες δεν ήταν πολύ για να τα ακούσουν αυτά. Παρακαλώ λοιπόν Λάβετε το υπόψη σας, κατά τον επόμενο προϋπολογισμό θα μας απασχολήσει και το θέμα αυτό ως πρόγραμμα πιλωτικό. Τρίτον, να σας πω ότι ίσως έχετε δει ότι η βιβλιοθήκη μας, η λιμπρερή μας κάνει πάντοτε πολύ ωραίες περιλήψεις επί διαφόρων θεμάτων. Πολύτιμες. Πολλές φορές δεν ξέρουμε τι κάνει η βιβλιοθήκη. Επιτελεί εξαιρετικό έργο. Και σας λέω, αν θέλετε κάποιο θέμα να το επεξεργαστείτε, δεν είναι ανάγκη να πάτε στην επιστημονική υπηρεσία, μπορείτε να απευθυνίσετε και στη βιβλιοθήκη μας, διότι η βιβλιοθήκη μας εξυπηρετεί και αυτό το σκοπό. Θα πάτε στο διαδίκτυο, θα δείτε τι προσφορά έχει η βιβλιοθήκη, εις ό,τι αφορά συνόψεις επιστημονικών θεμάτων που μας έχουν απασχολήσει. Πολύ ε, χρήσιμο αυτό. Ε, όταν θέλετε να ε, μιλήσετε για διάφορα θέματα. Αυτά είχα να σας πω και τώρα πάμε στο σημείο 8 της ημερήσιας διάταξης. Ε, θαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρση των εμποδίων στα δικαιώματα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο συντάκτης είναι ο Μόρτεν Λόκεγκαρτ και του δίνω αμέσως το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Το θέμα που θα μας απασχολήσει για το πώς μπορούμε να προωθήσουμε αυτά τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών είναι πάρα πολύ επίκαιρο γιατί πρέπει να αποδείξουμε στους πολίτες μας ποια είναι η αξία της δουλειάς μας. Η έκθεση από την περσινή χρονιά ε, κατέληγε σε κάποιες συγκεκριμένες συστάσεις για το πού πρέπει να δράσουμε και νομίζω ότι αυτό αποτελούσε και την κατάλληλη αφετηρία για τις προσπαθίες μας. Αυτό το οποίο είναι πιο σημαντικό για εμένα είναι πως έχουν, μάλλον χαίρουν ε, πάρα πολλών δικαιωμάτων οι Ευρωπαίοι πολίτες, χωρίς όμως να τα γνωρίζουν. Και αυτό αποτελεί και το πρόβλημα. Μία από τις προτάσεις που κάνω στις παραγράφους 1 και 2 της ανακοίνωσης είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών κάτι το οποίο προσπαθώ να πετύχω με το κείμενο στο πρώτο άρθρο. Για να γίνει με ένα συντονισμένο και δομημένο τρόπο, χρειάζεται λοιπόν να ακολουθήσουμε συγκεκριμένη στρατηγική και πρέπει να συνεργαστούν στο θέμα αυτό και τα διάφορα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό λοιπόν το έχω συμπεριλάβει και στο πρώτο άρθρο. Έχουμε και τη διοργανική ε, ομάδα η οποία θα συνεδριάσει μάλιστα σήμερα βρίσκεται στη δεύτερη παράγραφο και ξέρετε πως αυτή η ομάδα δεν ε, τα πάει και τόσο καλά για να το πω ευγενικά. Πρέπει λοιπόν να συνεργαζόμαστε καλύτερα στην ομάδα αυτή και το τονίζω με το συγκεκριμένο κείμενο. Περνώντας ε, στο πακέτο για την ελευθερία των ΜΜΕ Αναφέρουμε εκεί στην, ε, στο δικαίωμα του να πληροφορείται κανείς από ανεξάρτητες πηγές. Είναι ένα θέμα ε, το οποίο πρέπει να σχολιάσουμε και για τα ΜΜΕ νομίζω η φωνή της Επιτροπής μας είναι σημαντική. Αρκεί λοιπόν να το συζητήσουμε εδώ και να το δρομολογήσουμε για την αναγνώριση των πτυχίων Παράγραφος 5. Περίοδη μελέτης και φίτησης σε άλλα κράτη-μέλη. Ε, νομίζω ότι για το θέμα της κινητικότητας υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες και ελπίζω πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει περισσότερες προσπάθειες. Θα σταματήσω εδώ και ε, θα αφήσω το λόγο στους υπόλοιπους συναδέλφους. Ευχαριστώ. Μαρία Θα είμαι πολύ σύντομη γιατί διάβαζα τώρα την ε, πρόταση που μας κάνει ο συνάδελφος και θα ήθελα από τα σημεία τα οποία έχει συμπεριλάβει στο σχέδιο γνωμοδότησης την προσπάθεια που θα πρέπει να καταβάλουμε για να έχουμε πιο καλούς μηχανισμούς για την αναγνώριση των ακαδημαϊκών πτυχίων και των περιόδων φίτηση σε άλλα κράτη-μέλη. Νομίζω είναι ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε διάφορα κράτη, όπως και εσείς και εγώ λαμβάνω πολύ συχνά καταγγελίες, ε, παράπονα και αναφορές από τους πολίτες ε, για θέματα παρόμοια. Νομίζω λοιπόν πως η ιδέα αυτή είναι εξαιρετική και το έχει τοποθετήσει στο σωστό σημείο. Wydaje mi się, że, że wartym jest podkreślenia fakt e, dotyczący e, prawa obywateli do... Νομίζω ότι πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι οι πολίτες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε δημόσια πληροφόρηση. Υπάρχουν πολλοί οργανισμοί που δεν έχουν ενιαίες διαδικασίες. Πιστεύω λοιπόν ότι καλό θα ήταν να αναδείξουμε περισσότερο το ζήτημα αυτό. Μέχρι τώρα δεν είχαμε χρόνο να μιλήσουμε για τις τροπολογίες στο κείμενο, αλλά αυτό το σημείο πρέπει να το υπογραμμίσουμε ότι χρειαζόμαστε απλουστευμένες και ενιαίες διαδικασίες στην πρόσβαση στην ενημέρωση. κυρία Παλιαδέλη. Απλώς στο σημείο 5 θα ήθελα να ρωτήσω τον συνάδελφο. Ε, την Επιτροπή, φαντάζομαι την Κομισιόν, να εντείνει τι προσπάθειες για την ανάπτυξη εργαλείων βελτίωση τη ακαδημαϊκής αναγνώριση. Αυτό είναι ένα ζήτημα που είχε απασχολήσει εδώ και χρόνια την Επιτροπή ε, μετά τη διαδικασία της Μπολόνια, από τη διαδικασία της Μπολόνια και τα Δεν καταλαβαίνω, δεν προσπαθώ να καταλάβω τι άλλα εργαλεία όταν ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της ε, ε, σύγκλησης αν θέλετε και της δυνατότητα ε, απασχόλησης προκύπτει από την εφαρμογή του στα κράτη-μέλη. Δηλαδή δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσε να κάνει η Επιτροπή. Θα ήθελα να μου εξηγήσετε τι εννοείται με, με αυτή τη διατύπωση. Ευχαριστώ. Äh, και εγώ θέλω να παρέμβω στη συζήτηση. Το σημείο 5 μου φαίνεται αδύναμο. Όπως είπε και η κυρία Παλιαδέλη, εδώ πάμε να τετραγωνίσουμε τον κύκλο, γιατί όχι... και στα πλαίσια της διαδικασίας της Μπολόνια αυτό είναι ένα ζήτημα που μπλοκάρεται από τις εθνικές κυβερνήσεις. Και σε μια χώρα όπως τη Γερμανία, μεταξύ ομοσπόνδων κρατηδίων υπάρχουν διαφορές. Αναγνωρίζομαι στον, στο ένα, όχι στο άλλο. Αυτή είναι η κατάσταση στην Ευρώπη. Αλλά αυτό δεν φτάνει. Δεν χρειάζεται μόνο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Χρειάζεται και σε άλλα επαγγέλματα κάτω από το επίπεδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των πτυχίων από εκεί. Κάπου λοιπόν στο κείμενο πρέπει να λέει ότι η δουλειά που κάνουμε, το έργο που επιτελούμε για τους πολίτες θα πρέπει να καταστεί περισσότερο ορατή. Αναφέρομαι στα κομμένιους, εράσμους, όλες τις ε, προσφορές εκπαίδευσης και προσφορές για τους νέους που έχουμε. Γιατί όλα αυτά είναι μέσα, είναι εργαλεία που στοχεύουν στους ε, πολίτες, στους νέους, στους ηλικιωμένους, στους μεσήλικες, ε, δηλαδή ε, εκπαιδευτικές προσφορές, προσφορές στα πλαίσια της κινητικότητας θα πρέπει να ενταχθούν επίσης σε αυτό το κείμενο, διότι έτσι θα προσελκύσουμε περισσότερο τους πολίτες από ό,τι με άλλα πράγματα. Πολίτες που έχουν παιδιά, που έχουν εγγόνια, ενδιαφέρονται πολύ για να αποκομίσουν τα καλύτερα ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης τα παιδιά και τα εγγόνια τους. Αυτό το σημείο 5 λοιπόν θα πρέπει να διευρυνθεί λίγο, να επεκταθεί, να γίνει καλύτερο. Δεν βλέπω να παρεμβαίνουν άλλοι. Οπότε αυτή ήταν μια πρώτη συζήτηση. Και... Ε, α, α, η Κομισιόν θέλει να πει τίποτα πριν ε, μιλήσει ο κύριος Λόκεγκάρτ. Ορίστε, Κομισιόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, θα κάνω θετικά και εγώ σχόλια από την πλευρά μου. Η Κομισιόν συμφωνεί με το γεγονό ότι οι πολίτε θα πρέπει να έχουν καλύτερη γνώση των δικαιωμάτων του και να είναι πραγματικά με, ε, να είναι Ευρωπαίοι πολίτε. Θα πρέπει να του χρησιμοποιήσουμε, συνειδητοποιήσουν ότι είναι πολίτε τη Ευρώπη. Επίση, εργαζόμαστε πάρα πολύ για να υπάρχει, υπάρχει μια πληροφόρηση, μια νέα πληροφόρηση όσον αφορά τους πολίτες αυτό. Όσον αφορά τους φοιτητές, δημοσιεύθηκε ένας οδηγός το 2010 για τους φοιτητές εντός ΕΕ και μέσα σε αυτήν προσπάθεια που γινόταν για τους νέους, ένα κίνημα που γινόταν και βεβαίως θα το συζητήσουμε σήμερα ε, μακρότερο επί του θέματος αυτού στα πλαίσια στην άλλη Επιτροπή, όπου θα υπάρχει το θέμα για την νεότητα και αυτό το πρόγραμμα θα δημιουργηθεί για να δημιουργηθεί ένα εργαστήριο ιδιαίτερα για τους νέους οι οποίοι θα πρέπει να μάθουν την κινητικότητα που υπάρχει εντός της ΕΕ και οι φοιτές ιδιαίτερα. Νομίζω για μας είναι κάτι το οποίο επιστηρίζουμε πλήρως και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμβολή της δικής σας Επιτροπής στην προσπάθεια που κάνουμε και εμείς με τη σειρά μας. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε μου για τη σχολεία σας. Και εγώ θα ήθελα να πω πως πιστεύω πως πραγματικά υπάρχει εδώ μια συνένεση θα λέγαμε για αυτό το θέμα αυτό και τους εταίρους οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια είναι σκοπός μας αυτή τη στιγμή να υπάρξει ένα αποτέλεσμα μετά από αυτή την εργαστή συνεργασία που υπάρχει μεταξύ μας. Λαμπρά, λέει η πρόεδρος. Ε, εντάξει, μέχρι τις 6.12, σύντομα δηλαδή, είναι, θα πρέπει να είναι... Ε, ε, ε, α, όχι, όχι, μισό λεπτό, μισό λεπτό, γιατί τον μπέρδεψα με την Πολόνη. Πιο νωρίς είναι ακόμα αυτή. Την επόμενη 28 ενδεκάτου είναι η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών. 28 ενδεκάτου. Οπότε να τηρήσετε αυτές τις προθεσμίες παρακαλώ. Πολύ σύντομα ο εισηγητής είναι οι σκιώδεις ελπίζω να προλάβουν. Αλλιώς πρέπει να δώσουμε παράταση της διαδικασίας και δεν ξέρω αν γίνεται. Το πρόβλημα είναι ότι η Επιτροπή Αναφορών είναι υπεύθυνη και στις 12 Ιανουαρίου ψηφίζουν, οπότε εμείς θα πρέπει νωρίτερα να έχουμε γνωμοδοτήσει. Καλά. Θα επιταχύνουμε λοιπόν αναγκαστικά. Ωραία, ευχαριστώ. Και πάμε στο σημείο 9, παρουσίαση μελέτης με θέμα ενθάρρυνση των ιδιωτικών επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα. Αλεξάνδρα Ούζελακ, συντονίστρια μελετών Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων. Είναι εδώ μαζί μας. παρακαλέσαμε την κυρία να μας κάνει μια μελέτη για το θέμα και χθε όλη μέρα μιλάγαμε για επενδύσεις στον πολιτισμό ιδιωτικές και δημόσιες και νομίζω ότι θα βοηθήσει και το έργο μας στα πλαίσια των επομένων προγραμμάτων που θα μας παρουσιαστούν σήμερα και παρακαλώ σε 15 λεπτά το πολύ να μας παρουσιάσει την εργασία της. Θα θυμάστε ότι είχαμε 2,6% του ΑΕΠ ε, προέρχεται από την πολιτιστική βιομηχανία των, ε, και, των, και τις τέχνες. Πρέπει όλα αυτά να επηρεάσουν λοιπόν την πολιτική και τα προγράμματά μας και πρέπει να δοθούν κίνητρα ώστε το Συμβούλιο Υπουργών να καταπιαστεί με τα θέματα αυτά πολύ σοβαρά. Ελπίζω η μελέτη να μας δώσει καινούργιες γνώσεις και περισσότερα συμπεράσματα. Η κυρία Ούζελακ έχει το λόγο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από εμάς πώς η ιδιωτική χρηματοδότηση μπορεί αυτή τη στιγμή να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς προσπαθούμε να δώσουμε μια καλύτερη και πλήρη γνώση για τα κίνητα τα οποία θα πρέπει να υπάρξουν για την χρηματοδότηση. Προσπαθήσαμε να εκφανίσουμε μια έκθεση η οποία περιλαμβάνει ερωτηματολόγιο για την έρευνα την οποία κάναμε. Αυτή η μελέτη λοιπόν ή έχει έρθει από την Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων, καθώ επίση από τη Λουμπλιάν, από το Σκέντρο για τη Διεθνή Σχέση, από τον κύριο Τσόπιτ, του Πανεπιστήμιου τη Λουμπλιάν. Το βασική έρευνα έχει γίνει από το Δεκέμβριο του 2010 και είχαμε βεβαίως ακροάσεις που γίνανε για το θέμα αυτό. Νομίζω αυτά είναι τα βασικά στοιχεία τα οποία ήθελα προκαταπολικά να υποβάλω. Η μελέτη προσπαθεί να δει τους διάφορους μορφές επενδύσεων που μπορεί να γίνει και ποια είναι εκείνα τα κίνητρα τα οποία έχουν και μπορούν να δοθούν. Στο δεύτερο κεφάλαιο προσπαθώ να δει τις γενικότερες τάσεις μέσα στην αψινόψη, όσον αφορά την ιδιωτική ε, χρηματοδότηση καθώς επίσης και τους μηχανισμούς οι οποίοι μπορούν να δώσουν περισσότερη όθηση και να δώσουν κίνητρα για τη χρηματοδότηση των μορφωτικών εκείνων εκδηλώσεων και ποια είναι τα εμπόδια τα οποία υπάρχουν. Επίσης γίνεται μία μικρή ανάλυση για τα τεκτογνώμενα στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο περιλέψει και αυτό μέσα στη μελέτη που υποβάλλουμε. Αυτή τη στιγμή η αντίληψη η οποία υπάρχει και τις νέες προοπτικές για τη βιωσιμότητα αυτών ε, δημιούργησε μια πίεση για την περαιτέρω χρηματοδότηση που θα πρέπει να έρχεται από άλλου τομεί. Υπάρχει όμω αυτή τη στιγμή μια έλλειψη για μια συστηματική ροή πληροφοριών η οποία θα πρέπει να γίνει σε αυτό το πένο. Δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία από τα ιδιωτική χρηματοδοτήσει για τα μολυτιστικά θέματα, ούτε υπάρχει μια μεθοδολογία συγκριτική η οποία μπορούσε να βοηθήσει πολύ τα πράγματα. Οι λεπτομέρειε βεβαίω είναι οι οποίες αναφέρουν πώς ακριβώς γίνονται τα πράγματα και στη μελέτη αυτή συμπεριλήφθησαν και στι μελέτες επίσης που έχουν γίνει από άλλες οργανώσεις σε άλλες χώρες. Ωστόσο τα, ωστόσο, τα υπαρχόμενα αυτή τη στοιχεία, επειδή έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορες μεθοδολογίες, είναι πάρα πολύ δύσκολο σήμερα να έχουμε μια συγκρισιμότητα αυτό το στοιχείο. Έτσι λοιπόν για τη μελέτη αυτή τα στοιχεία εκείνα τα οποία ε, έχουμε κάνει εμείς είναι ένα ερωτηματιολόγιο που στείλαμε στους υπουργού πολιτισμού των διαφόρων χωρών Επίσης υπάρχουν ερωτήσεις οι οποίες έχουν, ε, έχουν γίνει από στα στοιχεία εκείνα τα οποία έχουμε συλλέξει μέχρι τούδε και βεβαίω όλα αυτά άπτονται το Υπουργείο Πολιτισμού των διαφόρων χωρών και αυτά τα στοιχεία α, Βεβαίω ε, τα δεύτερα στοιχεία αυτά έρχονται από το Υπουργείο των Οικονομικών των διαφορών χωρών. Επίση, προσπαθήσαμε να κάνουμε ένα ολόκληρο συμπίλημα το οποίο θα είχε όλε αυτέ τι οργανώσει, οι οποίε περιλαμβάνονται μέσα και οι οποίε συμβάλλουν σε αυτό το τομέα μέσα σε αυτή τη μελέτη που έχουμε αναχείραση. Θα ήθελα αυτή τη στιγμή να σα πω πάρα πολύ σύντομα ποιε είναι εκείνε οι ιδέε, τα κόνσεπτ εκείνα τα οποία συνεπάρχουν. Ξέρετε, ο πολιτισμός και τα πολιτιστικά είναι ένας τομέας, είναι ένας που, ε, ε, ο οποίος έχει μεγάλη επίδραση και στον οικονομικό αλλά και ιδιαίτερα στον κοινωνικό τομέα, διότι άπτεται των πολιτιστικών εκείνων συμβάντων και γεγονότων και είναι πολύ ποικίλα αυτά για να υποτιμήσει κανείς θα πρέπει να εκτιμήσει την πολιτισμό σαν ένα ιδιωτικό αλλά και ένα εμπορεύσιμο είδο. Είδος. Έτσι λοιπόν οι πολιτικές στην Ευρώπη θα πρέπει έχουν ήδη μία δημόσια προσβασιμότητα και υπάρχει μία, ε, ένα, τα κείμενα τα, έχουμε, τα οποία έχουμε αναχείρα δικαιολογούν αυτή την αιτιολόγηση που σας έκανα. Υπάρχει οικονομική, κοινωνική, αλλά και ε, πολιτισμική, που είναι το πρώτο ε, αξία όλων αυτών των συμβάντων. Βεβαίω υπάρχει μια πολιτισμική βιομηχανία, θα λέγαμε των και νομίζω πως περιλαμβάνει ε, όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται για την κοινωνική ένταξη των καλλιτεχνών. Σκοπό τη το έχουμε αυτή τη στιγμή, το οποίο το, το αποδεικνύουμε μέσα από τη μελέτη μα, είναι μια μεικτή χρηματοδότηση που γίνεται δημόσιο και ιδιωτικού τομέα και προσπαθούμε να εστιάσουμε πολύ περισσότερο στην έμεση οικονομική υποστήριξη η οποία γίνεται και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να εξασφαλίσουμε ένα τέτοιο κόντεξ, πλαίσιο, το οποίο πραγματικά θα υπάρξει και περισσότερη η ιδιωτική αυτή υποστήριξη. Με όλα αυτά τα, δράματα ε, μπορούν να υπάρχουν προγράμματα τα οποία μπορεί να είναι πάρα πολύ εποφελία και των χωρών αλλά και ιδιαίτερα των κοινωνιών των διαφόρων μελών μας. Η ιδιωτική λοιπόν, έτσι όπως ε, η ιδιωτική επένδυση, έτσι όπως αυτή τη στιγμή αναφέρεται μέσα στην έκθεση είναι από τα άτομα, από τις επιχειρήσεις, από τις αιρές και όχι από δημόσιους οργανισμούς. Έτσι λοιπόν σκοπός αυτή τη στιγμή για την υποστήριξη είναι, είναι άμεσες επενδύσεις, χορηγίες, μεγάλες χορηγίες που εξασφαλίζουν τα έσοδα. Επίσης υπάρχει μια... Όλες αυτές οι πληρωμές οι οποίε γίνονται ε, καθοδηγούνται από διάφορου τρόπου. δηλαδή ποιο είναι το κέρδο το οποίο θα επιφέρουν, ποιο είναι το κοινωνικό όφελο το οποίο θα δημιουργηθεί και επίσης μέσω της αγοράς η οποία πραγματικά στηρίζει αυτά τα πολιτισμικά ε, συμβάντα, αυτά τα γεγονότα. Θα ήθελα πά, να σας δώσω μερικά βασικά στοιχεία, κλειδιά, αυτή τη Βασικά είναι ε, προσανατολισμένη αυτή η προσπάθεια προς την κρατική στήριξη βεβαίω. και υπάρχει μια πολιτική απόφαση η οποία χρειάζεται στα πλαίσια αυτά και υπάρχει αυτή. Επίσης υπάρχει μια ανάγκη ε, μεταρρύθμισε αυτό το τομέα για να γίνει πιο βιώσιμο, αλλά η πράξη αυτή τη στιγμή δείχνει η πρακτική ότι υπάρχουν ε, διάφοροι τομείς η προσπάθεια δημόσια γίνεται πολύ περισσότερο αυτή τη στιγμή για την υποστήριξη όλων εκείνων των, προσ... των ε, πολιτισμικών γεγονότων τα οποία είναι απόψεως της προμήθειας που γίνεται, δηλαδή της, της προσφοράς που γίνεται και υπάρχει ε, μία συμβολή των πολιτισμικών εκείνων οργανώσεων τα οποία πρέπει να επιδείξουν τα δυνατότητα του οποία για να ανάπτυξη αυτών των διαστηριοτήτων. Οι άμεσες επίσης προσπάθειες οι οποίες γίνονται, αλλά όλες αυτές απογειώνουν αν θέλετε την προσπάθεια καθώς επίσης οργανώσεις και τα και που συμμετέχουν, και όλες αυτές θα πρέπει περαιτέρω να διαφημιστούν αλλά και να προωθηθούν. Εάν δούμε πραγματικά ε, τη χορηγή η οποία γίνεται, αυτά έχουν μία μεγάλη σημαντική θα λέγαμε επίδραση, αν και αποτελούν μικρό ποσοστό. Σε πολλές χώρες υπάρχουν τα τα, οι χορηγίες οι οποίες έρχονται από τα παίγνια και από τον ΟΠΑΠ θα λέγαμε τον ελληνικό και, και βεβαίως αυτό το θέμα της δημόσιας υποστήριξης και χορηγίας είναι, είναι αφισβητούμενο καθότι σε περίοδους κρίσης μειώνεται. Επίσης θα πρέπει να, δοθούμε, να δούμε το θέμα πώς μπορεί να γίνεται μεταξύ κρατικής και ιδιωτικής επένδυση αυτούς τους τομείς το, το, σε αυτό τον τομέα το πολιτιστικό. Επίσης, θα πρέπει ε, ο ιδιωτικός τομέας να υπάρχει, να συμβάλλει, αλλά όχι να υποκαταστά πλήρως τη δημόσια χρηματοδότηση. Επίσης, οι οργανώσεις αυτή τη στιγμή που υπάρχουν ε, εταιρικέ και άλλες δημιουργούν ε, ένα, μια γέφυρα μεταξύ των καλλιτεχνών αλλά και της ε, επαγγελματικής δραστηριότητας τις οποίες αναπτύξουν. Υπάρχουν μελέτες οι οποίες γίνονται αυτό το θέμα, αλλά βλέπουμε ότι συστηματικά αυτά τα δύο δεν είναι συνδεδεμένα με ταξίδιους. Αφετέρου, το γεγονός ότι γίνει πιο επαγγελματικό η συλλογή ε, χορηγιών, η συλλογή κεφαλαίων για αυτό το θέμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή να χρησιμοποιηθούν αυτοί όλοι οι οι, συμμετέ, μετέχοντες για να υπάρξει περισσότερη συγκέντρωση χρημάτων για τέτοιες πολιτισμικές δραστηριότητε. Επίσης κάναμε τη συγκρίση μεταξύ τη Ευρώπης και Αμερικής και υπάρχουν τεράστιες διαφορές όσον αφορά τους προσανατολισμούς καθώς επίσης και τα αποτελέσματα συστήματα εντελώς διαφορετικά όσον αφορά και τα ποσά αλλά και τη δομή Ξέρετε υπάρχουν άλλα πολιτικά, άλλα νομικά καθεστώτα σε αυτές τις δύο πλευρές του Ατλαντικού και υπάρχει ε, διαφορά επίσης όσον αφορά την παράδοση που υπάρχει στις δύο αυτές τις πλευρές του Ατλαντικού. Ωστόσο, η παρούσα κοινωνική κρίση έχει, έχει μεγαλύτερη επίπτωση στην τέχνη από ό,τι αλλού. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο πιστεύουμε ότι η τέχνη και η καλλιτέχνη είναι αυτοί οι οποίοι πρέπει το περισσότερο και νομίζω πραγματικά βασικό σκόπος για την Ευρώπη είναι να υποστηρίξει την τέχνη και τους καλλιτέχνες σαν ένα δημόσιο αγαθό το οποίο υπάρχει και αυτό θα αποτελέσει ένα, ένα κίνητρο. Ε, νομίζω ποιε είναι αυτές οι οποίες δεν είναι οι ατέλειες οι οποίες υπάρχουν μεταξύ ιδιαίτερα για τις ε, πολιτισμικές εκείνες εταιρείες και τους προσανατολισμούς τους. Σε μια μικρή οικονομία όπου υπάρχουν υποστηρίξει εκ μέρου του δημοσίου καθώ επίση και του ιδιωτικού τομέα, τομέα Στην πρώτη ε, φάση χρειάζεται περισσότερη υποστήριξη που θα πρέπει να υπάρξει μεταξύ της δημόσιας ακρόασης αυτών των γεγονότων, καθώς επίσης και τις προσπάθειες που γίνεται των ιδιωτικών τομέων για την επεξήγηση των κολτόρων. Υπάρχει μια ολόκληρη σειρά συστάσεων τις οποίες κάνουμε αυτή τη στιγμή και θα αφήσω να φέρω μερικά από αυτά και ποιες είναι αυτές οι συστάσεις που, που σας κάνουμε είναι ανάπτυξη μια ισορροπία μεταξύ άμεση και έμεση δημόσια υποστήριξη, μια μεθοδολογία και ανάπτυξη όσον αφορά για την ε, συγκριτική πληροφόρηση, ανάπτυξη μια σταθερής ε, σταθερής δημόσιας υποστήριξης για να υπάρξει περισσότερη σταθερότητα, για να υπάρξει δημόσιο χαρακτήρα όσον αφορά του πολιτισμικού. Η δημόσια υποστήριξη είναι πολύ σημαντική. Ένα άλλο να υπάρχει μια ανάπτυξη της μεθοδολογίας για τη συλλογή συγκριτικών πληροφοριών. Πιστεύω πως αυτό Αυτό θα πρέπει να γίνει διότι μέχρι στιγμή υπήρχαν έλλειψη στοιχείων όσον αφορά τον, τον ιδιωτικό τομέα επένδυσης. Οι στατιστικές λοιπόν θα πρέπει να συγκεντρωθούν σε ένα συμπίλημα που θα πρέπει να γίνει για να λάβουν υπόψη τις ανάγκες ε, ε, ε, δημοσιοποίησης και προώθησης τέτοιων συγκριτικών πληροφοριών. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει μια συλλογή όσον αφορά τους φόρους οι οποίοι δημιουργούνται και ποιοι είναι οι κανονισμοί οι οποίοι διέπουν αυτή την, τους κανονισμούς. Επίσης ανάπτυξη τη υποστήριξη για την διεθνής οργανισμούς εκείνη και την, την παρακολούθηση των συγκριτικών στοιχείων και πρακτικών. Θα πρέπει εφόσον υπάρχει αυτή τη στιγμή επαγγελματοποίηση όσον αφορά τα θέματα αυτά, θα πρέπει και οι στρατηγικές που ακολουθούνται να είναι αντίστοιχες. Μία άλλη σύσταση είναι ε, θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη γνώση όσον αφορά τη φορολόγηση αυτών των θεμάτων για να υπάρχει προώθηση της ιδιωτικής ε, πρωτοβουλίας Επίσης, τα διάφορα μέτρα τα οποία είναι αυτή τη στιγμή, τα οποία υπάρχουν για τα κίνητα στον φορολογικό τομέα. Οι πολιτικές εκείνες που ασχολούνται στο φορολογικό για να υπάρξει μια ανάλυση συγκριτική όσον αφορά τις διάφορες χώρες για να, βρεθεί βελ, βρεθούν οι, οι βέλτιστες λύσεις. Το τελευταία σύσταση είναι οι διάφορες πολιτισμικές δραστηριότητες οι οποίες θα γίνονται από τις διάφορες αξίες πολιτισμικές οι οποίες σε κάθε χώρα. Πιστεύουμε πως και αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Πιστεύουμε ότι η προκλήση αυτή τη στιγμή είναι να υπάρχουν τέτοιοι μηχανισμοί στην κοινωνική πολιτική σε ένα τέτοιο οικονομικό περιβάλλον το οποίο ζούμε. Θα πρέπει να αναπτυχθούν οι αρμοδιότητες επίως χρειάζονται στον ιδιωτικό τομέα για την περαιτέρω ανάπτυξη των πολιτισμικών αυτών παρεμβάσεων και θα πρέπει να υπάρξει επίσης ένα νομοθετικό έργο το οποίο θα πρέπει να είναι ε, κατάλληλο για να υπάρξει βιωσιμότητα στον τομέα αυτό. Προσπάθησα να είμαι πάρα πολύ σύντομη. Έδωσα πραγματικά τα βασικά στοιχεία και περιμένω τις ερωτήσεις σας θα ήθελα να σας πω ακόμη, οι σε αυτή την έκθεση θα ήταν πάρα πολύ ευτυχεί να δεχτούν τα σχόλιά σα γραπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λάβαμε το έγγραφο από πλευρά σα και νομίζω ότι μπορούμε να το διαβάσουμε, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ε, οποιαδήποτε στιγμή κριθεί απαραίτητο, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να ξεκινήσει και μια μικρή συζήτηση για τις προτάσεις σας, για τα ευρήματά σας ε, θα δώσω λοιπόν πρώτα στη Μαρία το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω καταρχήν την ε, ε, εισηγήτρια για μια έκθεση η οποία μου φάνηκε εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Και το πρόβλημα είναι να βρει κανείς έγκυρες πληροφορίες που να απογράφουν πραγματικά την κατάσταση στα διάφορα κράτη-μέλη. Εμένα μου αρέσει να μελετώ το θέμα αυτό και έρχομαι πολύ συχνά στη συζήτηση για τη σχέση μεταξύ ε, οικονομικών ε, συμφερόντων και πολιτιστικού κλάδου ε, που, έχω, που δημιουργεί προβλήματα γιατί τα στοιχεία του 2008 λένε για 3% του ΑΕΠ. Το 2009 ήταν το 1,7% και σήμερα μου λέτε ότι είναι το 2,5% του ΑΕΠ. Άρα λοιπόν λείπουν στοιχεία και είναι δύσκολο να ενημερωθεί κανείς για το πώς έχει πραγματικά η κατάσταση με τον ε, κλάδο του πολιτισμού σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Αυτό που θα χρειαζόμαστε θα ήταν ένα είδος ΣΔΙΤ, δηλαδή συμπράξη δημοσίου και ιδιωτικού ε, τομέα, έτσι ώστε να φέρουμε τα αποθητά αποτελέσματα. Θα ήθελα να εστιάσετε και στη διαφορά μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί ξέρουμε πως σε επίπεδο πολιτιστικών εκδηλώσεων στι Ηνωμένε Πολιτείες είχαν μια πιο ισχυρή τάση για χορηγίε, για επειδή υπήρχαν και τα φορολογικά πλεονεκτήματα. Ίσως λοιπόν θα μπορούσατε να εξηγήσετε καλύτερα ποια είναι η διαφορά, ποια είναι η ουσιαστική διαφορά μεταξύ των όσων γίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες στηρίξανε οι ιδιώτες περισσότερο τον πολιτισμό. Γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το σημείο οι επιδόσεις μας ακόμα δεν είναι εξαιρετικά ε, φιλόδοξες. Συλλέγουμε τώρα ερωτήσεις, θα απαντήσετε μετά, θα δώσω το λόγο και στους άλλους συναδέλφους. Ο κύριος Φίσας. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι πολύ ικανοποιημένο από το γεγονός πως έχουμε αυτό το έγγραφο το οποίο ζήτησα από την αρμόδια υπηρεσία στην αρχή της θητείας μας μέσω της πολιτικής ομάδας και μετά μέσα της επιτροπής μας γιατί ε, είναι πολύ χρήσιμη. Υπήρχε πραγματική ανάγκη για μια τέτοια μελέτη ε, και μπορούμε όλοι να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία. Ε, πρόσφατα είδα μια περίληψη, μια σύνοψη που μου έστειλαν και νομίζω καλύπτει όλα τα σημεία τα οποία υπάρχουν ε, και τα οποία εγώ θεώρησα πως θα ήταν ενδιαφέρον να συζητήσουμε. Κάτι επιπλέον, γιατί νομίζω ότι το μοναδικό σχόλιο που θα μπορούσα να κάνω είναι για την συγκριτική μελέτη που χρειάζεται να γίνει μεταξύ ε, Ευρωπαϊκής, κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, δεν ε, συμπεριλάβατε χώρες όπως η Γερμανία, όπως η Γαλλία, που είναι σημαντικές, γιατί ήταν η Πολωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Δανία κτλ. Δεν σας λέω γιατί δεν συγκρίνατε με την Ισπανία, γιατί σε καμία ισπανική κυβέρνηση, δυστυχώς μέχρι σήμερα, ούτε αριστερή, αριστερών ε, πεπεθήσεων, ούτε δεξιών δεν είχαμε κάτι τέτοιο. Ένα από τα σημεία στα οποία θα ήθελα επίσης να επιμείνω είναι αυτά τα οποία έθιξε και η συνάδελφος Μαρία. Δηλαδή τη σύγκριση που πρέπει να γίνει μεταξύ του ευρωπαϊκού συστήματος και του αμερικανικού. Γιατί πάντα είμαστε, αν θέλετε, ναι, ζηλεύουμε, ζηλεύουμε όχι μόνο στον πολιτισμό αλλά και στον αθλητισμό τις επιδόσεις που έχουν σε επίπεδο χορηγιών οι ΗΠΑ. Ίσως θα έπρεπε να δούμε στο νομοθετικό πλαίσιο εκεί ε, τι προσφέρει. Και βέβαια σε συνθήκες κρίσης δυστυχώς όλα τα θέματα αυτά αντιμετωπίζουν περικοπές στις επενδύσεις στον πολιτισμό για παράδειγμα και νομίζω και στον αθλητισμό συμβαίνει κάτι αντίστοιχο. Καλό θα ήταν λοιπόν αυτές τις δημόσιες επενδύσεις οι οποίες δεν θα πρέπει να εξαφανιστούν και εγώ πιστεύω πως πρέπει να έχουμε ένα μεικτό σύστημα πώς θα μπορούσαμε όμως να σταθμιστούν αυτές οι περικοπές με χορηγίες από τους ιδιώτες. Γιατί δεν μπορούμε να αφήσουμε το θέμα του πολιτισμού στους ε, ιδιώτε. δεν μπορούμε να του πούμε κάντε μας τη χάρη, στηρίξτε ε, τον αθλητισμό και, τον πολιτισμό. Όχι, θα πρέπει να τους δώσουμε κάποια πλεονεκτήματα, ίσως κάποιες φορολογικές ελαφρύνσεις, που θα τους οδηγήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Μήπως λοιπόν κάποιοι ευρωπαϊκοί νόμοι πρέπει να αλλάξουν και να βελτιωθούν. Ευχαριστώ για την παρουσίαση και τις συστάσεις. Μιλήσατε για εναρμόνιση μέτρων ΦΠΑ χωρίς να θίγεται το ιδιαίτερο καθεστώς των αγαθών αυτών. Την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο ψηφίσαμε για την μείωση των ΦΠΑ για ψηφιακά πολιτιστικά αγαθά και υπηρεσίες. Τι γνώμη έχετε εσείς γι' αυτό, γι' αυτό το πολιτικό μέτρο και πώς ορίζετε εσείς τις πολιτιστικές υπηρεσίες γιατί και αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Τι ακριβώς καλύπτεται όταν μιλάτε για πολιτιστικές υπηρεσίες που τις αναφέρατε. Και επίσης ε, η τελευταία σας σύσταση ε, αφορούσε ε, δράσεις στην πολιτική για τον πολιτισμό που θα διέπεται από διαφορετικές αξίες πολιτιστικές. Τι ακριβώς εννοείται, γιατί δεν το κατάλαβα και πολύ καλά. Ευχαριστώ, κύριος Μπόρης. Δύο ερωτήσεις σε σχέση με το κύριο θέμα μας. Πρώτη ερώτηση. Το ποσοστό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα του πολιτισμού. Ξέρουμε καλά ότι υπάρχουν πολλά κονδύλια για την υποστήριξη της καινοτόμου δύναμης και της προώθησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εννοείται ότι τα διατιθέμενα κονδύλια δεν δημιουργούν εμπόδια γιατί είναι χαμηλά τα κατόφλια, τα ανώτατα, τα ανώτατα όρια, με συγχωρείτε. Ε, πιστεύετε ότι με ευρωπαϊκά κονδύλια θα μπορούσαν όλα αυτά να προωθηθούν αποτελεσματικότερα. Δεύτερη ερώτηση αφορά τον κινηματογράφο. Δεν ξέρω αν έχετε επεκτείνει την έρευνά σας και εκεί, αλλά στις Ηνωμένε Πολιτείε λειτουργεί ο ιδιωτικός τομέας με αρκετή επιτυχία. Στην Ευρώπη, κατά κανόνα, ε, χρησιμοποιούμε κρατικά κονδύλια και ο ιδιωτικός τομέας ε, κατά μικρό ποσοστό χρηματοδοτεί την κινηματογραφία. Βλέπετε εδώ κάποια εμπόδια, γιατί δεν συμμετέχει δηλαδή περισσότερο ο ιδιωτικός τομέας. Η αγορά είναι τεράστια. Και νομίζω ότι θα μπορούσαμε εδώ να αξιοποιήσουμε το ευρωπαϊκό δυναμικό, που και αυτό είναι τεράστιο. γιατί το ιδιωτικό κεφάλαιο δεν ε, συμμετέχει σε αυτές τις δραστηριότητες. Ευχαριστώ και εγώ θα έκανα αυτή την ερώτηση, οπότε περιτεύει να παρέμβω. Ε, ποιος θα απαντήσει εσείς, οι συνάδελφοι. Ναι, δεν ξέρω. Όχι, όχι, α, όχι, α, α παρανόηση. Νομίζω ότι ήταν και άλλοι συναδελφοί σας εδώ μαζί. Η αλλαγή είχε να κάνει με την διαφορά μεταξύ των, ε, του ευρωπαϊκού και του αμερικανικού συστήματος. Ξέρετε, η φορολογική μεταρρύθμιση έλαβε χώρα στις πολιτείες στο τέλος της δεκαετίας του 60 και εκεί υπάρχουν πολύ περισσότερα φορολογικά πλεονεκτήματα τα οποία είναι πιο περίπλοκα, περισσότερο ξεκάθαρα και στην μελέτη αφιερώσαμε όσο χρόνο μπορούσαμε στο θέμα αυτό. Αυτές οι φορολογικές ελαφρύνσεις εκεί είναι υψηλότερες από ό,τι είναι στην Ευρώπη. Και θεωρούμε πως όταν κάποιος φορολογούμενος φορολογείται πολύ, θεωρεί πως έχει εκτελέσει τα καθήκοντά του ενώπιον του πολιτισμού και δεν δίνονται κίνητρα για να στηρίξει κανείς παραπάνω. Στις Ηνωμένε Πολιτείε η κατάσταση αποδεικνύει πως ο κλάδος του πολιτισμού δεν είναι ιδιαίτερα σταθερός. Δηλαδή υπάρχει μια μακριά παράδοση που δίνει φορολογικές ελαφρύνσεις σε όσους κάνουν χορηγίες και στους δωρητές Οπότε και εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται μία μελέτη με περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί βέβαια εμείς δεν είχαμε χρόνο ούτε χώρο για να αφιερώσουμε ε, πολλές προσπάθειες στο θέμα αυτό. Αυτό που κάναμε ήταν είναι να κάνουμε μια περιγραφή των γενικότερων τάσεων. Στο παράρτημα της μελέτης δίνουμε περισσότερες λεπτομέρειες για το σύστημα στις Ηνωμένε Πολιτείες και κάνουμε και μια απογραφή των φορολογικών μέτρων που θεωρούμε ότι αποτελούν κίνητρο για τέτοιου είδους ε, συμπεριφορά. Ε, τα μέτρα αυτά είναι διασπαρμένα σε διαφορετικούς νόμους ε, στην Ευρώπη και γι' αυτό ο κλάδος του πολιτισμού δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά, γιατί πολλές φορές δεν γνωρίζουν καν την ύπαρξή τους. Σε μία από τις συστάσεις προτείνουμε να κάνουμε και μία κατηγοριοποίηση αυτών των φορολογικών ελαφρύνσεων ε, γιατί διαφορετικά ε, οι πληροφορίες αυτές μπορεί κανείς να τις βρει μεν αλλά ο τρόπος με τους οποίους παρέχονται δεν είναι ιδιαίτερα φιλικός προς το χρήστη. Οπότε ναι, χρειάζεται ένας κατάλογος για τα φορολογικά συστήματα στην Ευρώπη και τα ε, πλεονεκτήματα που προσφέρουν σε ανθρώπους που κάνουν δωρεές ή χορηγίες. Είναι σημαντικό λοιπόν να έχει κανείς μια επισκόπηση συστηματική της κατάστασης στην Ευρώπη. Ένα είδος ανθολογίας, για παράδειγμα, ή ένα έργο που θα χαρτογραφήσει και θα παρακολουθήσει τις εξελίξεις ε, ενός θέματος που είναι και περίπλοκο και όπως αναλαμβάνω υπάρχει μεγάλη διασπορά ε, σε διάφορα νόμους και στα διάφορα κράτη ε, υπάρχουν και αποκλήσεις έτσι ώστε οι δικαιούχοι να γνωρίζουν τι ακριβώς μπορούν να κάνουν. Χρειάζεται λοιπόν να προωθήσουμε και την κουλτούρα της προσφοράς αλλά και της κουλτούρας της Απόδοση αυτή τη προσφορά, γιατί πιστεύω ότι οι ιδιωτικέ εταιρείε και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να στηριχθούν, να παίξουν το ρόλο που μπορούν και να προσελκυθούν σε αυτήν την κοινή πλατφόρμα και βέβαια χρειαζόμαστε και στοιχεία τα οποία θα έχουμε με πιο συστηματικό τρόπο και που θα ακολουθεί παρόμοιες μεθοδολογίες. γιατί βεβαίω τα εθνικά περιβάλλοντα στα διάφορα κρατημέλη είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. για αυτή τη μελέτη, ε, την περιπτωσιολογική μελέτη, να σα πω πω η Ευρώπη είναι πολύ διαφορετική μεταξύ της. Και μπορούσαμε όντως να έχουμε επιλέξει οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα. Εμεί προσπαθήσαμε απλώ να επιλέξουμε τελείω διαφορετικέ πραγματικότητε, όχι μόνο τις καλέ περιπτώσεις, αλλά και αυτές τι οποίες δεν λειτουργεί το σύστημα, γιατί βεβαίω θέλουμε να έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα βοηθήσει όλους. Ανακαλύψαμε πως το Ηνωμένο Βασίλειο και οι κάτω χώρες έχουν συστήματα που έχουν τα πιο προχωρημένα μέτρα και εκεί είναι και ε, ορατές οι πολιτικές που ακολουθούνται. Επίσης εκεί οι επιχειρήσεις και οι ε, ενώσεις οι πολιτιστικές συνεισφέρουν πολύ στα όσα γίνονται και πιστεύουμε πως για τις χώρες αυτές υπάρχουν και πολλά στοιχεία. Δεν επιλέξαμε τη Γαλλία, ίσως γιατί δεν είχαμε κάποιο γαλλόφωνο, ερευνητή γαλλόφωνο στην ομάδα μας. Όταν αξιολογούμε ε, τέτοια στοιχεία, οι πηγές μας ε, είναι σε διαφορετικές γλώσσες. Οπότε επιλέξαμε να εστιάσουμε σε χώρες της γλώσσας στην οποία μιλάμε, έτσι ώστε να μπορούμε πρώτο χέρι να μάθουμε τι γίνεται, γιατί δεν είχαμε μεταφραστές. Πιστεύουμε πως αυτό το οποίο παρουσιάσαμε είναι αρκετά αντιπροσωπευτικό της ευρωπαϊκής πραγματικότητας. Ηνωμένο Βασίλειο, Πολωνία, κάτω χώρες, Σλοβενία, Πολωνία, Σλοβενία είναι νέα κράτη-μέλη. Θέλαμε να δούμε πώς λοιπόν αυτοί οι εισερχόμενοι ανταποκρίνονται στις προκλήσεις, αν υπάρχουν βασικές διαφορές, πώς μπορούν να ξεπεραστούν. Η Ιταλία είναι χώρα της Μεσογείου, για αυτή την επιλέξαμε. Και εκεί θεωρούσαμε ότι η κατάσταση είναι αρκετά ε, διαφορετική. Για την εναμόνιση του ΦΠΑ, Ψάξαμε παραδείγματα. Είχαμε και νομικό στην ομάδα μας που παρακολούθησε το θύμα, το θέμα, με συγχωρείτε. Η εναρμόνιση γίνεται με κάποιες συνεχιζόμενες εξαιρέσεις οι οποίες αποδεικνύουν ε, και τα θετικά αποτελέσματα της εναρμόνισης. Δηλαδή το να πιέσουμε προς αυτή την κατεύθυνση για μας είναι σημαντικό, είναι ένα καλό επιχείρημα, αλλά θα θέλαμε να συνεχιστούν αυτές οι εξαιρέσεις, γιατί και πάλι ο πολιτισμός μπορεί να θεωρηθεί και ως προϊόν κοινή ωφελία. Και δεν είναι εύκολο να συρριχθεί ο πολιτισμός μόνο σε ιδιωτικά κεφάλαια. Ίσως λοιπόν κάποιο είδους ε, χορηγίες ή επιχορηγήσεις για τις πολιτιστικές ομάδες και ενώσεις. Αυτό ε, θεωρήθηκε θέμα σημαντικό για το οποίο δεν μπορούμε να δώσουμε μια εύκολη απάντηση. δεν ξέρουμε πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Πάντως η μελέτη αποδεικνύει πως ε, χρειάζεται έρευνα στο θέμα της φορολογικής πολιτικής εδώ και πιστεύουμε ότι κάποιος θα πρέπει να αναλάβει αυτή τη μελέτη γιατί υπάρχουν ε, πολλές ερωτήσεις και αυτές που κάνατε που άπτονται του θέματος της φορολογίας. για τις διαφορετικές αξίες του πολιτισμού. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να βλέπουμε τον πολιτισμό ως αγαθό, εμπορεύσιμο. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει και κοινωνικές επιπτώσεις. Επιτρέψτε μου να σας διαβάσω τα σχετικά από την έκθεση. θα πρέπει να το αξιολογούμε με ολιστικό τρόπο. Όχι μόνο δηλαδή ε, να εξετάσουμε τα οικονομικά ωφέλη που προσφέρει, αλλά και τα κοινωνικοπολιτιστικά πλεονεκτήματα. Αυτό είναι τμήμα των συστάσεων, γιατί θέλουμε αυτές οι πτυχές να τονιστούν Και γι' αυτό πιστεύουμε πως θα πρέπει να έχουμε αυτό το μείγμα της μικτής χρηματοδότησης. Ο πολιτισμός έχει διάφορες αξίες τις οποίες εμείς θα πρέπει και να διατηρήσουμε και να προωθήσουμε. Κύριε Ράτιμορ, θέλετε να λάβετε το λόγο, έχετε σηκώσει το χέρι σας. Ξέρετε, εμείς σε αυτά τα πλαίσια μπορούμε να κάνουμε κάτι σαν μια πρόταση, μια αίτηση προς την Κομισιόν, γιατί το χαρακτηριστικό αυτό που υπάρχει εδώ και βεβαίως θα ήθελα να ακούσω τις συντάξεις σας. Μιλάω σαν Ιταλός και μιλάω όμως σαν Νότιος Ευρωπαίος κατά αρκετά νομίζω ότι οι περισσότερες αυτές οι ιδιωτικές παρεμβάσεις γίνονται περισσότερο για την διαφήμιση και όχι τόσο για φορολογικούς λόγους. Αυτό περιλαμβάνει κινδύνους καθότι εάν πάρετε πραγματικά το κείμενο ενός φεστιβάλ ή οτιδήποτε υπήρχουν εκεί γεμάτο σύμβολα που έρχονται πραγματικά από διάφορες οργανώσεις, από διάφορες εταιρείες που κάνουν αυτή τη χορήγηση. Στην Αμερική όμως υπάρχουν μειώσει φορολογική και αυτοί οι μειώσει πληρώνουν για τα μουσεία, τι βιβλιοθήκε κλπ. Και υπάρχουν επίση πρωτοβουλίε οι οποίε σιγά σιγά γίνονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε μπορούν να πάνε προς τον χορηγό ο οποίος έχει κάποια ωφέλη από αυτό. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πάρουμε και να συγκρίνουμε μερικά αποτελέσματα από αυτή τη προσπάθεια και κατά αυτόν τον τρόπο να καλέσουμε την ΕΕ ή τα οργανώσεις ΕΕ να κάνουν μία μείωση όσον αφορά την φορολογική μείωση τέτοιου είδου πολιτισμικών εκδηλώσεων. Κατά αυτόν τον τρόπο πραγματικά νομίζω μπορούμε να συμβάλλουμε εμείς για ότι σε, ό, σε χώρες έτσι έχουν τα πράγματα όπως σας είπα και ας πρέπει να καταλάβουμε πως μέσα αυτή την έκθεση μπορεί να υπάρχουν συστάσεις οι οποίες μπορεί να είναι χρήσιμες και μπορούμε βεβαίως κατά τον τρόπο να ανοίξουμε το έβρος αυτής της προσπάθειας η οποία γίνεται και πιστεύω πως η δική μας Επιτροπή κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί να δώσει μια περισσότερη όθηση σε αυτή την προσπάθεια που μπορεί να γίνει στον τομέα αυτό. Αγαπητέ μου κύριε Ράτιμο, δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα η κυρία. Εμείς αναθέσαμε αυτή τη μελέτη και το τι θα κάνουμε εμείς θα το αποφασίσουμε μετά. Να διαβάσουμε τη μελέτη, να δούμε τι συμπεράσματα θα βγάλουμε και αυτό θα είναι η βάση για το έργο μας το επόμενο διάστημα για τις ε, πολιτιστικές βιομηχανίες ότι σήμερα η συζήτηση θα περιορίζεται σε αυτή τη μελέτη. Εμένα θα με ενδιέφερε και θεωρώ ότι είναι πολύ καλό να γίνει μια έρευνα και για τις βόρειες, τις σκανδιναβικές χώρες. Οι Σουηδοί έχουν δυσκολίες χρηματοδότησης του κλάδου του πολιτισμού. Οπότε θα είχε νόημα να δούμε πώς χρηματοδοτείται ο πολιτισμός ε, ε, στις βόρειες χώρες. Ε, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θεωρώ ότι είναι βόρεια σκανδιναβική χώρα. Ε, ίσως δεν υπήρχε αρκετή χρηματοδότηση για να διευρύνετε τη μελέτη σας και ως προς τη Γαλλία κλπ. Γιατί είναι σημαντική χώρα. Μας ενδιαφέρει όμως, δεν σας κατηγορώ δηλαδή για το εύρος της μελέτης, αλλά θέλουμε να πάρουμε πολλά στοιχεία, πολλά περισσότερα για να δούμε που βρίσκονται οι διαφορές. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν πολλές. Αν πάρετε το Ηνωμένο Βασίλειο, ας πούμε, την Ολλανδία, τη Σλοβενία, την Πολωνία, ε, δεν είμαι βέβαιη αν αυτές οι χώρες δίνουν μια καλή εικόνα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές χώρες που πρέπει να μελετηθούν, ίσως στα πλαίσια μιας επόμενης μελέτης και όταν θα διατίθενται τα απαραίτητα κονδύλια. Θέλετε να απαντήσετε κάτι. Ναι, για τις, ε, για τους, τις χορηγίες... Βεβαίως πρέπει να προωθούνται ε, η χορηγία αποσκοπεί και σε ίδιο όφελος, προαγωγή, πρόθεση κλπ. Οπότε οι χορηγίες περιορίζονται σε πολύ μεγάλες ορατές εκδηλώσεις ε, έγκριτων πολιτιστικών οργανισμών, ενώ άλλοι δεν θα έβρισκαν τόσο εύκολα ε, χρηματοδότηση από χορηγούς. Ε, ίσως τα τραπεζικά ιδρύματα όπως στην Ιταλία θα μπορούσαν να παίξουν ρόλο ε, κάτι που να υπάρχει δηλαδή όχι αποκλειστικά ως όφελο στην ατζέντα τους, αλλά και ως κοινωνική, κοινωνικό αντίκτυπο. Βεβαίως ε, η επιλογή που κάναμε έγινε και δεν ε, ανατρέπεται, αλλά από την άλλη πρόκειται για ένα πρώτο βήμα. Η πρώτη αυτή έρευνα έχει μία αξία, αλλά για να έχουμε πιο συστηματική και συνεχιζ... Ε, για να έχουμε καλύτερη ενημέρωση και ε, ένα input στην πολιτική χρειάζεται μία συνεχιζόμενη έρευνα. Και οι εθνικές έρευνες που συμπεριλαμβάνουν και γνωρίζουν όλα τα προβλήματα εν προκειμένου θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε ένα ε, εγχειρίδιο, αν θέλετε, μια συλλογή των πολιτικών σε έναν τόμο που θα ενημερώνεται. Αν θέλει κανείς να καταπιαστεί με τη μέθοδο της αλλαγής και της βελτίωσης του ιδιωτικού τομέα στην πολιτική, χρειάζεται κάτι τέτοιο για να παρακολουθείτε την κατάσταση εν εξελίξη και να στηρίζετε τις αποφάσεις σας πάντοτε σε ενημερωμένα στοιχεία. Μάλιστα, θα πρέπει λοιπόν να γίνουν και περιπτωσιολογικές μελέτες και έρευνες όπως αυτή και σε άλλες χώρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εργασία σας. Δώσατε φρέσκα στοιχεία που θα τα αξιοποιήσουμε. Ευχαριστώ. Πάμε. Α, μήπως η Κομισιόν θέλει να πει κάτι. Υπάρχει κάποιος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κυρία Σαμπρόν, θέλετε να προσθέσετε κάτι. Δεν είναι και απαραίτητο δηλαδή, αν δεν ε, επιθυμείτε. Ω κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα πρώτα να σα ευχαριστήσω και να πω και να συμφωνήσω μαζί σας σε σχέση με την παρατηρήση που οποία κάνατε για τη σημασία που έχει αυτή τη στιγμή να υπάρχουν ομάδες οι οποίες αντικατα αντικατοπτρεύουν την κατάσταση. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την παρουσίαση αυτή της έκθεσης όσον αφορά την ιδιωτική επένδυση στον τομέα των πολιτισμικό, καθότι φρονούμε πως στην καταρχήν αυτή η προσπάθεια πάει συνάδει με την προσπάθεια που κάνουμε και εμείς για τη χρηματοδότηση του πολιτιστικού τομέα και επίσης συμπίπτει με την υιοθέτηση του προγράμματος για το για τη δημιουργική Ευρώπη την οποία αυτές τις μέρες περνάμε. Κατά αυτόν τον τρόπο έχουμε αντιμετωπίσει τη δυνατότητα να υπάρχει ένα νέο εργαλείο χρηματοδότησης για την δημιουργία και τον πολιτιστικό τομέα. Αυτό το εργαλείο θα, θα υπάρχει σε λίγο, όσον ούπο. Αυτό είναι σε εκπόνηση βεβαίως αυτή τη στιγμή, υπό εκπόνηση και ασπαζόμαθα την ανάλυση η οποία έχει γίνει μέσα σε αυτά τα πλαίσια, δηλαδή την ανυπαρξία των συγκριτικών στοιχείων. εργαζόμαθα βέβαια για να τα προκτήσουμε αυτά, προσπαθούμε να οθήσουμε το Συμβούλιο και συνεργαζόμαστε με τη Γενική Διεύθυνση Περιοχών επί των θεμάτων αυτών για τη χρηματοδότηση. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ μπορώ να σας ζητήσω να σκεφτείτε και εσείς εκ μέρους Κομισιόν που για τη χρησιμοποίηση ε, της δικής σας, ε, ε, του δικού σας τμήματος της έρευνας για να υπάρξει ένα follow-up ε, για αυτή την προσπάθεια η οποία έχει γίνει, για αυτή την έρευνα, τη μελέτη. Γιατί ξέρετε υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση η οποία γίνεται για αυτό το θέμα και το δικό αυτή τη στιγμή το department, ε, το τμήμα των ε, ερευνών είναι πάρα πολύ σημαντικό και μπορεί να συμβάλλει τα μάλα σε αυτή την προσπάθεια. Και νομίζω μακροπρόθεσμο μπορεί να βοηθηθεί πολύ αυτό το πράγμα για το δικό σας τμήμα της έρευνας. Θα χαρούμε ιδιαιτέρως εάν έχουμε αποτελέσματα, διότι πραγματικά υπάρχουν χρήματα που σας διατίθενται για αυτό το τομέα και μπορούτε να έχετε και λαμπρά αποτελέσματα τα οποία θα μας επιφέρουν καλά αποτελέσματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία. Σημείο 10. Ο κύριος Μπερλιγκουέρ θα μας ε, παρουσιάσει την έκθεση για την Πολόνια. Δεν θα πω πολλά, την περασμένη φορά είπα τα πολλά. Σας δίνω αμέσως το λόγο. Κύριε Μπερλιγκουέρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα και εγώ να επαναλάβω στην παρουσίαση μου η οποία γίνεται στην προηγούμενη παρουσίαση που είχε γίνει και νομίζω πως θα ήταν ένα μου σήμερα να επαναλάβω τα ίδια. Ωστόσο θα επιμείνω σε μερικές πτυχές η οποία είναι πολιτική σημασία, υψή της πολιτικής σημασίας από τη δική μας πλευρά που εξετάζουμε την έκθεση αυτό. Λαμβάνοντας βέβαια υπόψη ότι οι συνάδελφοι είχαν το κείμενο, έχουν το κείμενο αναχείρας για αυτή την πρόταση την οποία έχω κάνει για την πρόταση ψηφίσματο και κατά αυτόν τον τρόπο είναι, έχουν μπει καλύτερα στο θέμα αυτό το οποίο εξετάζουμε και του όλου της όλης θεματολογίας. Πιστεύω πραγματικά το βασικό πράγμα το πολιτικό το οποίο θα πρέπει επίσης να κάνουμε με, σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με, με την Ολομέλεια βεβαίως πώς μπορεί πραγματικά αυτή η απόφαση να περάσει από την Ολομέλεια και να είναι μια σταθερή, μια μόνιμη απόφαση που θα ληφθεί και αυτό θα σημαίνει ότι μια τέτοια απόφαση είναι, σκοπός είναι να υπογραμμιστεί ο ρόλος τον οποίο έχουν οι ευρωπαϊκές όργανα όσον αφορά την οικοδόμηση της, του ευρωπαϊκού χώρου της ανώτερης εκπαίδευσης. Φαίνεται ότι είναι μοναδικό αυτή τη στιγμή ότι σε αυτό το επίπεδο ε, όλες οι αρμοδιότητες αν θέλετε είναι των κρατών μελών ενώ αυτή τη στιγμή έχουμε ένα χώρο ευρωπαϊκό της ανώτερης εκπαίδευση, ο οποίο δεν είναι συντονισμένο αυτό το πούμε καθαρά και παστρικά και πεντακάθαρα ότι έτσι έχουν αυτά τα πράγματα πολύ λοιπόν στο ε, Βασιλείου και Βεβαίω είναι ένα άλλο θέμα το οποίο επίση θα επανέλθουν πάλι και πολλοί σε αυτό το, το κοινοβούλιο για αυτό το θέμα. Αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο φρονώ πω θα ήθελα εγώ να επιμείνω και να παραμείνω στη Λισαβόνα. Άρθρο 55 της ε, Λισαβόνο, το οποίο λέει αυτή τη στιγμή θα πρέπει να υπάρχει μια ποιοτική εκπαίδευση θα συμβάλλει όλο και περισσότερο αλλά και θα ε, βοηθήσει τα κράτη-μέλη σε μεγαλύτερη συνεργασία σε αυτό το πράγμα. Το λέει λοιπόν πάρα πολύ σαφό. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι εναλλακτική λύση, κάτι φλού το οποίο δεν υπάρχει. Είναι σαφές μέσα στο κείμενο της Λισαβόνος και διευκρινίζω ότι ενθαρρύνοντας τη συνεργασία και προσπαθώντας αυτή τη στιγμή όλο να συμπληρώσει, να ε, προάγει την προσπάθεια και κατά αυτόν τον τρόπο να αναπτυχθεί, να αναπτυχθεί η ευρωπαϊκή διάσταση της ανώτερης έκδοσης. Βλέπετε μας λοιπόν σε δίκη υπάρχει μια ευρωπαϊκή αυτή η διάσταση που σας είπα για, τις για να υπάρχει μια κινητικότητα των φοιτητών και των καθηγητών, καθώς επίσης και μια αμοιβαία αναγνώριση όσον αφορά τα πτυχίων τα οποία, ε, τα οποία έχουν αποκτηθεί σε μια ξένη χώρα. Αυτή είναι η διαδικασία της Μπολόνιας. Και βεβαίως έδωσε την εντολή στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σύμφωνα με τις νομοθετικές διαδικασίες τι ε, κανονικές, να υπάρξει ένας κανονισμός αυτό είναι ο τίτλο το οποίο υπάρχει κατά σε αυτό το κεφάλαιο και εμεί νομίζω πραγματικά, ε, αν ξεκινήσουμε έτσι, είμαστε εντό των πλαισίων τη συνθήκη. Και βεβαίω μπορεί αυτό να επιγίνει ένα, να πάρει τη μορφή ενό νόμου. Στην ανακοίνωση λοιπόν των κομισών βλέπω μια ενθάρρυνση η οποία υπάρχει, καθώ επίση επανέρχομαι και λέγω ότι το καινοτόμο κοινό σημείο είναι ότι μεταξύ πολιτικού και Κοινοβουλίου υπάρχει μια σύγκριση όσον αφορά αυτή την όθηση η οποία πρέπει να γίνει προς τα μπρος. Και λέγεται εδώ ότι όλη η προσπάθεια της ανωτέρας εκπαίδευση ε, ε, ανήκει στα κράτη-μέλη, ωστόσο στα πλαίσια της αυτής της ε, διαδικασίας Μπολόνιας, ότι τόσο η έρευνα όσο αναφορά την έρευνα, όσο και τις οποιασδήποτε σπουδές οι οποίες γίνονται περαιτέρω από αυτό, ε, συμβάλλουν περισσότερο σε μια ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και ότι ξεπερνάνε τα σύνορα και δεν παίρνουν ενό των κρατών μελών. Έτσι λοιπόν θα πρέπει, ξέρετε υπάρχει ένας ολόκληρος μεγάλος κατάλογος εδώ πραγμάτων τα οποία αναφέρονται και αυτό σημαίνει πραγματικά ότι εμείς έχουμε μια αρμοδιότητα για να επιλύσουμε αυτό το θέμα. Και επίσης λοιπόν θα πρέπει αυτή τη στιγμή να τολμήσουμε πολύ περισσότερο από αυτό που έχουμε κάνει μέχρι τούδο, διότι η προσπάθεια τη Μπολόνια έχει εφαρμοστεί σε ορισμένε χώρες μόνο. Ένα άλλο πιο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι ότι υπάρχει μια διαφορά μεταξύ ε, και κίνδυνο της Ευρώπης. Υπάρχει μια ανισορροπία θα λέγαμε όσον αφορά την εφαρμογή της αυτής της, ε, της προσπάθειας η οποία ε, θα πρέπει και οι μεν και οι δε να καταλάβουν ότι είμαστε Ευρωπαίοι, ότι όχι μόνο υπάρχει ένα spread και εδώ, διότι ξέρετε αυτό το spread <laughs> το οποίο οικονομικός παράγοντας, ξέρετε πάρα πολύ καλά τι κακό κάνει αυτό το spread. Έτσι λοιπόν θα προπαρεύουμε και σε σχέση για αυτή την, και συγχωρήστε με για αυτή την, την παρομοίωση την οποία κάνουμε τα οικονομικά, διότι αυτή η ανισορροπία πραγματικά ε, ε, ασκεί κυρώσει εναντίον εκείνων των φοιτητών οι οποίοι έρχονται από αυτέ τι χώρε και ότι βρίσκονται πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία να συνεργαστούν, να ενταχθούν ε, μέσα στις υπόλοιπε χώρε τη Ευρώπη. Εφόσον πραγματικά, για παράδειγμα, υπάρξει μία ανεχρώση των τίτλων και υπάρχει μεγαλύτερη κινητικότητα, νομίζω πραγματικά αυτά θα πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα, τα παιδιά εκείνα τα οποία έρχονται από πουδήποτε της Ευρώπης. Έτσι λοιπόν, ποια είναι η αρμοδιότητα όσον αφορά την εξέβριση αυτής της ε, ισορροπίας και ποια είναι εκείνα τα οποία πραγματικά μπορούν να συμβάλλουν για να υπάρξουν αυτά τα μέτρα τα οποία μπορούμε να οδηγηθήσουμε σε αυτό το θέμα. Θα πρέπει να δούμε ότι υπάρχουν δύο μονοπάτια τα οποία ακολουθούνται καθότι αυτή τη στιγμή υπήρξε ένας αποκλεισμό ε, ε, αντικοινοτικός όσον αφορά τη, αυτή τις προσπάθειες της Μπολόνιας, τα οποία πραγματικά ακολουθήκαν από τα κράτη-μέλη, με ένα τέτοιο τρόπο όπου οι διετής αυτές προσπάθειες που γίνονται μεταξύ των Υπουργών ε, Πολιτισμού ή εκπαίδευση σε αυτό το θέμα, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία κάνανε ήταν εκτός ε, έψιλον. Και πιστεύω πραγματικά θα, ε, θα πρέπει να αλλάξει, διότι δεν θα θέλω πραγματικά αυτή τη στιγμή να πω στις λεπτομέρειες, διότι θα σκούραζα πάρα πολύ. Το Συμβούλιο και η Κομισιόν λοιπόν αυτή τη στιγμή μαζί με εμά πρέπει να κληθούν να διορθώσουν αυτή τη διαδικασία. Διότι στη στιγμή εκείνη τη στιγμή που υπάρχει μια συνάντηση η οποία γίνεται πίσω το Συμβούλιο της Ευρώπης και όχι εκτός της Ευρώπης θα πρέπει να είναι τα κράτη-μέλη εκείνα τα οποία συμμετέχουν διότι μερικέ φορέ πραγματικά συνέρχονται και υπάρχει μια soft συνάντηση η οποία γίνεται και η οποία τάχα μου δεν εντάσσεται στα πλαίσια της ΕΕ. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα πρέπει να γίνονται στα πλαίσια της ΕΕ για να υπάρχουν και όλα εκείνα τα πλαίσια πλεονεκτήματα τα οποία προκύπτουν. Και αφετέρου υπάρχει νομική βάση η οποία προκύπτει από τις συμφωνίες οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ΕΕ. Και νομίζω πραγματικά δεν πρέπει εγώ σαν Ιθαελός να κάνω μόνο το δικηγόρο εδώ και να τον αγορηθεί για αυτά τα θέματα. Αλλά πρέπει και οι Πολωνοί και οι Δανέζοι και οι υπόλοιποι θα πρέπει να αναλάβουν και αυτή την προσπάθεια και την πρωτοβουλία να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια. Δεύτερη παρατήρηση την οποία θέλω να κάνω εξή. Εμεί θέσαμε, θα ήταν υπενθυμίσω στου συναδέλφου στην πρότασή μα το εξή, ότι το στόχο τη αποτελεσματικότητα στο, στο ευρωπαϊκό χώρο μετά τη διαδικασία της Πολώνης ήταν στο σκοπό να να υπάρξει μία διαφοροποίηση των διαφόρων στοιχείων που υπάρχουν σε κάθε χώρα, αλλά παράλληλα να υπάρχει αυτή τη στιγμή η δυνατότητα κινητικότητα εντό εψηλών ΕΕ. Κινητικότητα. Αυτό είναι η πιο βασική λέξη και πρέπει να δούμε ποια είναι τα αποτελέσματα αυτή τη προσπάθεια. Και θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει όχι μία θεωρητική, μη συγκεκριμένη, αλλά πώ στην πρακτική αυτό ο τίτλο μπορεί να είναι έχει αξία να μπορεί να αναγνωρίζεται και πιστεύω πως αυτή τη στιγμή ότι η Ιταλία επειδή είναι ένα τίτλο, αν θέλετε ένα τίπλωμα, ότι αυτό το τίτλο με αυτό το τίτλο, με αυτό το πτυχίο να μπορεί να πάει στη Γερμανία, Γαλλία ή αλλού στην Ευρώπη και ότι με αυτό το, το πτυχίο ε, μπορεί να εργαστεί ή να έχει τις δυνατότητες που έχει. Αυτό το πρόβλημα το οποίο δεν έχει επιληθεί είναι εγενές πρόβλημα της προσπάθειας οι οποια έχει ξεκινήσει και βεβαίως κατά αυτόν τον τρόπο πιστεύω πως αν το ξεπεράσουμε αυτό μπορεί να υπάρξει ε, μια, καλύτερος, ε, μια καλύτερη αποτίμηση όσον αφορά τις ε, αποκτηθήσεις γνώσεις μέσω ενός πτυχίου στη χώρα που έχουν γίνει. Ένας ερευνητής το πραγματικά, ο οποίο σέβεται τον εαυτό δεν μπορεί να το κάνει μόνο στη χώρα του. Αυτό είναι γελίο. Πραγματικά τα πράγματα, οι πληροφορίες αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν παγκοσμίω. Νομίζω γυρίζουν γύρω-γύρω μας. Αυτό είναι ο ρόλο ε, και ποιο είναι το αποτέλεσμα το αυτό, ότι αυτή τη στιγμή τα πανεπιστήμια μα είναι κλειστά, είναι εθνικά, δεν έχουν γίνει παγκόσμια, δεν έχουν αποκτήσει μια διάσταση ευρωπαϊκή. Και πραγματικά δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να επιβάλλουμε στου νέου μα αυτού τι συνθήκε οι οποίοι πραγματικά είναι ξεπερισμένοι. Ακόμη δύο παρατηρήσει τι οποίε θα ήθελα να κάνω. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο σήμερα είναι ένα θέμα κοινωνικό το οποίο ανακύπτει. Και σε αυτό το τομέα, σε μερικέ χώρε υπάρχουν μερικοί ε, φοιτητέ οι οποίοι ε, αποκλείονται γιατί είναι πολύ ακριβά τα πανεπιστήμια και αυτό είναι μια ζημία η οποία γίνεται, μια χασούρα διότι για το 2020 η Λισαβόνα είχε προβλέψει κάτι άλλο από αυτό. Μέσα από τη Λισαβόνα λοιπόν και μέσα από τη διαδικασία της Λισαβόνας θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Δεύτερη παρατήρηση που θέλει αφορώ το εξή. Εγώ είχα την δυνατότητα να έρθω σε επαφή του με τους φοιτικές συλλόγους και φοιτητέ ακόμη οι οποίοι ε, μόνοι του ε, σπουδάζουν σε ξένα παραπιστευμένα. Ή, ξέρετε, οι φοιτητέ είναι απόντες. Αυτή ξερετε οι φοιτητε ειναι απόντε. αυτη η οποία υπάρχει και η οποία είναι διακυβερνητική δεν μπορεί να βασιστεί στο γεγονός ότι η διδακτική διαδικασία αυτή τη στιγμή θα είναι στο κέντρο της προσπάθειας. Μπορεί να κάνει τη μεταρρύθμιση, δεν μπορεί να κάνει αυτή την αλλαγή με τα learning centers που είναι μια πολύ βασική αλλαγή η οποία γίνεται στην καθημερινή μας ζωή και στη διδακτική μας. Έχουμε εμείς, έχουμε μια διδακτική διαδικασία η οποία έχει ε, βάση με τη διδασκαλία και τις εξετάσεις. Αλλά σήμερα θα πρέπει ο φοιτητή θα πρέπει να συμμετέχει ενεργώς σε αυτή την προσπάθεια της εκπαίδευσης, της εκπαίδευσης σε όλη την προσπάθεια, σε όλο και μερικά πανεπιστήμια, μερικά ε, χώρες έχουν βελτιώσει αυτή τη στιγμή. Αλλά όταν όταν γραφόταν οι, οι όπερες παλαιότερα ε, γραφόταν πάνω στις παρτιτούρες μόνο Ιταλικά, Αντάντε, Αντάτζο κλπ. Πιστεύω ότι υπήρχε μια διεθνοποίηση δηλαδή τότε, ενώ σήμερα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτή το, ε, το, το μέτρο, συνοδευτικό μέτρο το οποίο θα πρέπει να υπάρχει για να βοηθάει. Το πρώτο βέβαια βήμα υπέρ το, το πίση και λέγω ε, σου δίνω τα λεφτά και εσύ είσαι στο φοιτητή στο εξωτερικό. Δεν θα ήταν πολύ πιο σωστό όπως το είπαν οι συνάδελφοι μου από το Μάστριχ να δώσουμε τα λεφτά στο πανεπιστήμιο που υποδέχεται. Εάν πάει κανείς από τη Ρώμη στο Παρίσι από το πανεπιστήμια ε, οι Παρισινοί θα πρέπει να είναι αυτοί οι οποίοι να έχουν την υποδομή για να δεχθούν τον Ιταλό φοιτητή και όχι να δώσουμε τα λεφτά στον Ιταλό φοιτητή για να πάει στο Παρίσι. Εφόσον πραγματικά το κάνουμε αυτό θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα το οποίο είναι ισορροπημένο και το οποίο θα είναι αναγνωρίσιμο κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν το Πανεπιστήμιο τη Σαπιέντσα αυτή τη στιγμή δεν δέχτηκε ένα φοιτητή ε, ε, που είχε κάνει τις σπουδάσεις του στις Ηνωμένες Πολιτείες διότι πραγματικά δεν είχε σπουδάσει ε, στη Σαπιέντσα. Και πώς λεγόταν αυτό το Αμερικάνικο, ήταν το, το MIT, Institute of Masters of Technology. Σκεφτείτε τι γίνεται. Βλέπετε αυτή τη στιγμή στην δίνω αυτά τα παραδείγματα τα οποία θα πρέπει να γίνουν να ε, συγγνώμη που αυτή τη στιγμή έχω πάθος και σας πήρα πολύ χρόνο, αλλά θα πρέπει να ρυθμιστούν αυτά τα θέματα, μια και καλή. Δεν πολλοί μένει πολύς χρόνος, 20 λεπτά έχουμε. Μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου, σε 10 μέρες δηλαδή, ε, λίγη η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών. Θα ψηφίσουμε τον Ιανουάριο και μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου πρέπει να έχουμε τις τροπολογίες. Να το έχετε υπόψη σας αυτό. Καλό καγκάρ. Θέλετε ο κύριος Ράκημα. Τώρα θα συζητήσουμε αυτό το θέμα. Και εγώ εξετά προτιμάζω τροπολογίες που θα τις υποβάλουν αυτό το χρόνο. Θέλω να υπογραμμίσω και άλλα σημεία μας τα οποία θα ενισχυθούν μέσα στην έκθεση. Είναι το θέμα δηλαδή της αναγνώρισης των διπλωμάτων. Ο ποιο σημείο ο προλαλής σας τα είπε πολύ σωστά, δεν είναι μόνο τα ε, ε, ε, ακαδημαϊκά πτυχία τα οποία, αλλά υπάρχουν όλα εκείνα τα διπλώματα, αν θέλετε, τα οποία είναι επαγγελματικά και άλλα τα οποία θα συμπεριληφθούν μέσα αυτή. Και νομίζω αυτό το θέμα είναι πολύ πιο περίπλοκο. Το θέμα των φοιτητών τώρα, ακούσοντας αυτά τα οποία είπε ο Μπερλιγκουέρ προηγουμένως, Πρέπει να διασφαλίσουμε ως πως οι φοιτητέ του Εράσμου που έρχονται στη Γαλλία για παράδειγμα ναι, πρέπει Πρέπει όμως πριν φτάσουμε σε αυτούς θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τους φοιτητέ που είναι στην ίδια μας της χώρας. Νομίζω ότι πραγματικά αυτά είναι συνδεδεμένα στην προηγούμενη φορά προσπάθησα να διατυπώσω κάτι πολύ σαφώ. Για την αναγνώριση των διπλωμάτων θα πρέπει να υπάρξει ένα, μια αναγνώριση των διαφόρων πανεπιστημίων όσον αφορά τα εργαλεία τα οποία έχουν. Διαρωτώμε δηλαδή κατά πόσο δεν υπάρχει ένα τρόπο να υπάρξουν κριτήρια μάστρη και για τα πανεπιστήμια. Να υπάρξουν ένα δίπλωμα το οποίο θα πρέπει να αναγνωρίζεται αυτομάτως σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τόσο της εκατό, τόσο της εκατό, το οποίο έρχεται από τον καθηγητή και κατά αυτόν τον τρόπο γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει. Ξέρετε ότι υπάρχουν ε, κολέγια, φοιτικές αιστείες κλπ. κλπ. Όλα αυτά συνδέονται πάρα πολύ με αυτά που είπατε προηγουμένως. Καθώς επίσης και με τους τίτλους που αναφέρεται τα διπλώματα στα, στις ανθρωπιστικές επιστήμες είναι κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σύντομα όμως, ε, δεν έχουμε πολύ χρόνο, σύντομη θα είμαι. Θα επαναλάβω, δεν θα επαναλάβω αυτά που είπαμε την περασμένη φορά, απλώς ένα θέμα θα τονίσω, το οποίο έχει συμπεριλάβει και ο κύριος Μπερλιγκουέρ ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο απόκτησης προσόντων και αναγνώρισης προσόντων. Δεν ξέρω, θα μας βοηθήσει και το ευρωπαϊκό και τα 27 εθνικά πλαίσια για την αναγνώριση των εκπαιδευτικών τίτλων. Θα βοηθήσει δηλαδή τη διαδικασία αναγνώριση αυτό το σύστημα γιατί έχουν τόσο διαφορετική ταξινόμηση και κατηγοριοποίηση στα κράτη-μέλη, που το γερμανικό αμπιτούρ μπορεί να μην συμπεριλαμβάνεται στη Γαλλία σε κανένα επίπεδο, σε άλλες χώρες ε, είναι του επίπεδου 4, υπάρχει αδιαφάνεια. Δεν έχω λύση να προσφέρω, αλλά θα πρέπει με σοβαρότητα να εξετάσουμε αν το πλαίσιο αναγνώρισης, τα 27 εθνικά πλαίσια συν το ευρωπαϊκό, είναι ο καλύτερος τρόπος που θα συμβάλλει στο να λύσουμε το πρόβλημα και να έχουμε συγκρίσιμα πτυχία και διπλώματα στην Ευρώπη. Ευχαριστώ, κυρία Κώστα. Σύντομα, παρακαλώ, η κυρία Κώστα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πιστεύω κύριος Μπέρλιγκορ μίλησε και έχει την αξία ότι πραγματικά είπε ότι υπεχρέεται περισσότερο θάρρος, κουράγιο να υπάρχει και νομίζω πραγματικά πως αυτό είναι ένα σημείο που πρέπει να το περάσουμε όλοι για να φτάσουμε σε αυτό το, την Ευρώπη την οποία θέλουμε, στα πλαίσια της Ελλάδας βέβαια, και βεβαίω δεν θα πρέπει να έχουμε μόνο αριθμητικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και εργαλεία τα οποία θα υπάρχουν. Θα πρέπει. Πιστεύω ότι ε, συμφωνούμε όλοι αυτή τη στιγμή ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ενίσχυση αυτού του χώρου του ευρωπαϊκού και νομίζω ότι πως υπάρχει νομική βάση για αυτά τα θέματα και θα πρέπει να πάμε ακόμη περισσότερο, ε, όλη η διαδικασία αυτή θα πρέπει να γίνει εντός εισαγωγικών, περισσότερο κοινοτική εντός εισαγωγικών. Και νομίζω πως πραγματικά το οποίο έγινε προηγουμένως ότι σε αυτούς τους υπουργούς οι οποίοι συνέρχονται για λόγους καθαρά διαδικαστικούς εκτός ΕΕ είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν μία ε, κατεύθυνση την οποία είπε ο κ. Μπελιγουέρ και την οποία να σπαζόμεθα. Επίσης πιστεύω ότι και θα ήθελα να το υπογραμμίσω ότι θα πρέπει να υπάρχουν επιστώσεις για την εκπαίδευση και για τις σπουδέ εκείνε εντό εισαγωγικών που γίνονται, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σπουδέ εντό εισαγωγικών, λέει ο Μιλήτρια. Και κατά αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να υπάρχει αναγνώριση όχι μόνο των οργανώσεων που, των φοιτητών που ασχολούνται με το Εράσμου ή που κάνουν τι ανταλλαγέ στα πλαίσια του Εράσμου, αλλά και άλλων φοιτητών οι οποίοι ανέφερα προλαλή σα. Κατά αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε πω αυτοί οι οποίοι δέχονται τις υπηρεσίες των αυτό πολύ σιγά το κάνουν στα πλαίσια μόνο του Εράσμου και, και δέχονται. Αυτό που μπορούμε εμείς λοιπόν να προτείνουμε για τους φοιτητικούς ενώνου να υπάρχουν ε, ομάδες υποδοχής για αυτά τα πράγματα και τρίτον οι ομάδες εκείνες, οι οργανώσεις εκείνες που ασχολούνται με αυτά τα θέματα είναι να υπάρχει όλες εκείνες οι υποτροφίες ε, επιχορηγήσεις οι οποίες γίνονται από χώρα σε χώρα, να υπάρχει ένα δυνατότητα ενός σημείου υποδεχής και αυτό να είναι γνήσια όταν γίνονται. Νομίζω πραγματικά αυτή η έκθεση έχει το υπέρ της ότι να δώσει στα κράτη-μέλη την οδηγία εκείνη για να υπάρχει μια ανταπόκριση μεταξύ τους και μία αμοιβαιότητα και να μην υπάρχει εκείνο το εμπόδιο το οποίο είχε με τούδε το οποίο ήταν μία ανοργανωσιά όσον αφορά την αμοιβαία κίνηση. Η μέγιστη δυσκολία αυτή τη στιγμή που υπάρχουν παρά την προσπάθεια της, της ε, Μπολόνιας είναι είναι η τριετής αυτή παραμονή για τις ανθρωπιστικές σπουδές οι οποίες γίνεται και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να επανέλθουμε και να το εξετάσουμε καλύτερα. Ευχαριστώ. Ο επόμενος αγορητής. Ευχαριστώ. Αυτό που πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα είναι η αναθεώρηση της διαδικασίας της Μπολόνια ως προς την στρατηγική Ευρώπη 2020 και η κινητικότητα ως βάση των μέτρων μας. Η διαδικασία της Μπολόνια εφαρμόστηκε ε, χάρη στις προσπάθειες, στις μεγάλες προσπάθειες που κατέβαλαν όλα τα πανεπιστήμια και τα Ιδρύματα Τριτροβάθμιας Εκπαίδευσης, γιατί όλοι φοβόντουσαν ότι θα έχαναν την αυτονομία τους, για την οποία έδωσαν μάχες προεκατοντάδων χωρών και η οποία αυτονομία ήταν το βασικό χαρακτηριστικό πολλών πανεπιστημίων. Και εγώ συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος Μπερλινγκουέρ που λέει ότι οι σπουδαστές φοιτητές πρέπει να είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας και εκείνοι θα πρέπει να μπορούν να επιλέξουν στα τρία, ε, των τριών επιπέδων που θα σπουδάσουν στην Ευρώπη. Κατόπιν συνομιλιών με πολλούς Πριτάνης πανεπιστημίων ανεδίθη ένα σημαντικό θέμα που αφορά την ποιότητα. Όταν πάρει κανείς το bachelor σε ένα πανεπιστήμιο, αυτό δεν σημαίνει καθόλου ότι ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ενός άλλου πανεπιστημίου. Δηλαδή θα πρέπει να παρακολουθήσουν πρόσθετα μαθήματα οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για να ανταποκριθούν στις ε, ποιοτικές απαιτήσεις και πρότυπα άλλων πανεπιστημίων. Γι' αυτό χρειάζονται αυτά τα πλαίσια επαγγελματικών προσόντων για να λάβουν υπόσψη μας τα κριτήρια τα οποία αφορούν κυρίως την ποιότητα. Αυτό είναι ένα θέμα που το τονίζουν οι Πρετάνης. Ευχαριστώ κυρία Βαλιαδέλη. Τα ίδια που είπα και την προηγούμενη φορά, αλλά με βάση όσα είπε πριν από λίγο ο κύριος Μπερλίνγκουερ, θεωρώ ότι πραγματικά η αναγνώριση των ε, πτυχίων είναι το πιο σημαντικό εργαλείο, όχι μόνο σε επίπεδο επαγγελματικό για τους νέους, αλλά και σε επίπεδο ιδεολογικό αν θέλετε, γιατί είναι μια απάντηση στην ουσία σε αυτή τη διαλυτική τάση που εμφανίζουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια και, και επειδή οι νέοι είναι αυτοί οι οποίοι θα συνεχίσουν ή θα ολοκληρώσουν τη διάλυση της Ευρωπαϊκής ε, Συνύπαρξης. Επομένω θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η δυνατότητα αναγνώρισης των τριών επιπέδων. Τώρα, πώς το επιβάλλουμε αυτό στην, ε, στα κράτη-μέλη. Ε, έρχομαι από μια χώρα που μόλις τελευταία ε, ένας καινούριος νόμος προσπαθεί να περάσει αυτή την τριμερή διαβάθμιση στα επίπεδα σπουδών και έχουμε πολλές αντιδράσεις από τους φοιτητές και από διδάσκοντες. Ωστόσο θεωρώ ότι αναρωτιέμαι αν υπάρχει κάποιος τρόπος ενός ευρωπαϊκού συστήματος πιστοποίησης αυτών των ε, πτυχίων όπως είναι για παράδειγμα η πιστοποίηση των ξένων γλωσσών. Στα γαλλικά είναι το δεν ξέρω τι, το, στα αγγλικά είναι το δεν ξέρω τι, τα γερμανικά. Μήπως τελικά, χωρίς να υπερβούμε τις δυσκολίες εφαρμογή ενό τέτοιου συστήματος σε όλη την Ευρώπη, πράγμα που ενδεχομένω θα θεωρούν να και ομογενοποίηση, να βρούμε έναν τρόπο, ένα σύστημα που θα μπορούσε να πιστοποιεί αυτές τις τρεις βαθμίδες σπουδών και θα είναι ένα είδο ευρωπαϊκού πτυχίου ή ε, διπλώματος αναγνώρισης ανεξάρτητα που θα προκύπτει εθελοντικά και ανεξάρτητα από τις δεσμεύσεις των εθνικών κρατών. Μήπως δηλαδή μπορούμε να βρούμε ένα τέτοιο σύστημα χωρίς να υπερβούμε τις αγγυλώσεις των εθνικών δυσκολιών. Ε, οι φοιτητέ αδιαφορούν για όλα αυτά τα πράγματα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σα. Πρώτον, γιατί είναι αντιμέτωποι με μια ανεργία, δεν μετέχουν δηλαδή. Το μόνο που του ενδιαφέρει είναι να αποκατασταθούν επαγγελματικά. Και δεύτερον, γιατί αμφισβητούν τις προθέσεις αυτών που χειρίζονται τις τύχες τους. Φοβούμε δηλαδή ότι είναι απογοητευμένοι από τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε οι μεγαλύτεροι τις ε, αγωνίες τους και το μέλλον τους. Ε, θεωρώ πολύ σημαντική την πρότασή σας για την άμεση σύνδεση της έρευνας και της διδασκαλίας και πρέπει να εμβαθύνουμε προς αυτή την κατεύθυνση, οργανώνοντας ίσως κοινέ δράσεις ανάμεσα στον ευρωπαϊκό χώρο για την ανώτατη εκπαίδευση και για τον Ευρωπαϊκό Χώρο για την Έρευνα, φέρνοντας αυτούς τους δύο οργανισμούς, ε, τις δύο συνθέσεις πιο κοντά. Και θα τελειώσω πολύ σύντομα λέγοντας ότι οι υποδομές είναι απαραίτητη προϋπόθεση για, την, ε, για τα πανεπιστήμια. Πρέπει να υποστηρίξουμε ως Ευρώπη οικονομικά τις υποδομές των πανεπιστήμιων όχι μόνο σε ερευνητικό ή διδακτικό επίπεδο αλλά ακόμη σε σχέση και με, τον, με το Εράσμους Θεωρώ πολύ σημαντικό η χώρα που υποδέχεται να παίρνει τα χρήματα προκειμένου να, ε, να ανταποκρίνεται στις απαιτήσει των φοιτητών παρά να τα παίρνουν τα, τα κράτη έθνη και να βρίσκονται αντιμέτωποι οι φοιτητέ με πάρα πολύ κακές συνθήκες ε, ε εγκατάστασης, ε, υποδοχής και, και συντονισμού. Ε, θα κάνω τις τροποποιήσεις στο κείμενο αυτό, το οποίο όμως θεωρώ πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό για να ξαναδούμε τη διαδικασία της Μπολόνιας στην επόμενη δεκαετία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και εγώ να κάνω δύο παρατηρήσεις. Βρίσκω την έκθεση καλή. Είχα κάνει και εγώ κάποτε μια παρόμοια. Ε, παρακαλώ να λάβει δύο-τρία πραγματάκια ακόμη ο κύριος Μπερλινγκουέρ για τα European Credit Points, τα διδακτικά μόρια δεν αναφέρεται τίποτα, που είναι μεγάλο πρόβλημα γιατί παίρνουν ένα μόριο ε, για το ίδιο πράγμα κάποιοι, άλλοι τρία ε, μόρια. Και αυτό είναι μια ανισότητα. Πρέπει να βρεθεί ευρωπαϊκή ρύθμιση. Οι διδακτικές μονάδες δηλαδή. Επίσης, ε, το bachelor στο σημείο 13 το αναφέρετε, λέτε ότι θα πρέπει να προσανατολίζονται περισσότερο τα bachelor στην αγορά εργασίας. Καλό είναι αυτό. Αλλά πρώτα πρέπει να αναγνωρίζονται τα bachelor, το πρώτο πτυχίο. Κάποιοι θέλουν να συνεχίσουν. Τα πτυχία bachelor ακόμα και στην ίδια χώρα δεν αναγνωρίζονται από όλα τα πανεπιστήμια. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν ένα κανονιστικό πλαίσιο ε, που να, ώστε να μπορεί να λειτουργεί και η διαδικασία της, της Μπολόνια. Αυτό. Και επίσης ε, το σημείο 3 πρέπει να τα αλλάξουμε για την δημιουργία μιας πραγματικής ευρωπαϊκής επανεπιστημιακής ηθαγένειας. Ούτε η ηθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουμε ε, ολοκληρώσει. Κάτι άλλο πρέπει να το πούμε αυτό, όχι ηθαγένεια. Τώρα, η Κομισιόν Θέλεις να παρέμεις για την Πολόνια. Όχι. Όχι. Τώρα μιλάμε για την Πολόνια. Δεν μπορείς να έχεις το λόγο λοιπόν. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποιος θα λάβει το λόγο. Ο κύριος Τάισεν. Ορίστε. Ευχαριστώ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος γιατί μας περιμένει η Επίτροπος εκτός αιθούσης. Είμαι πεπισμένος πως η έκθεση αυτή αποτελεί μια εξωτερική ε, συμβολή στην Υπουργική για την Πολώνια του χρόνου τον Απρίλιο. Τονίζει τα θέματα που μας απασχολούν και τα διαστρωτικά αλλά και τα θέματα της ε, ύλη που διδάσκεται ε, και βεβαίως συνδέεται ε, με, τις, ε, το πλαίσιο ε, των ευρωπαϊκών δεξιοτήτων. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε όλα αυτά τα θέματα σε όλη τους τη διάσταση. Για τα κοινά πτυχία νομίζω πως θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα παγοθραυστικό το οποίο θα επιτρέψει μεγαλύτερη συνεργασία σε αυτό το επίπεδο μεταξύ κρατών μελών. Και ίσως θα έπρεπε να επιμείνουμε στη σχέση μεταξύ των πανεπιστημίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων για τα διδακτορικά, όχι μόνο τα ακαδημαϊκά διδακτορικά αλλά και τα βιομηχανικά διδακτορικά τα οποία έχουμε προωθήσει εμείς με τόση θέρμη για να βελτιώσουμε και να μεγιστοποιήσουμε την ε, τις επιπτώσεις αυτής της έκθεσης, νομίζω πως θα πρέπει να στείλουμε συγκεκριμένα αιτήματα στην Υπουργική που θα γίνει στο Βουκουρέστι του χρόνου και θα πρέπει να ζητήσουμε να ορίσουν ένα φιλόδοξο στόχο για την κινητικότητα των φοιτητών και να εστιάσουν στις βασικές, στις βασικ... στα βασικά εμπόδια, για παράδειγμα, του κατά πόσο κανείς μπορεί να μεταφέρει ένα φοιτητικό δάνειο έτσι ώστε να το πληρώνεται σε μια ξένη χώρα. Όπως επίσης και το θέμα της πανεπιστημιακής ύλη ε, που θα μας επέτρεπε αν είχαμε κοινή ύλη να ξεπεράσουμε τα προβλήματα της αναγνώρισης. Τώρα, θα πρέπει να δούμε πόσο διάφανες είναι οι εκθέσεις για αυτά που έχουμε μέχρι σήμερα για την διαδικασία τη Μπολόνια δεν είναι ευανάγνωστα. Θα πρέπει να είναι πιο εύκολη η πρόσβαση και από του φοιτητέ και από του πανεπιστημονιακούς για να ξέρουν σε ποιο σημείο τη όλη διαδικασία είναι το δικό του σύστημα. Θα χρησιμοποιηθεί λοιπόν αυτή η διαδικασία υποβολή εκθέσεων ω ένα όπλο για καλύτερη και πιο εναρμονισμένη εφαρμογή τη διαδικασία τη Μπολόνια σε όλη την ευρωπαϊκή ε, επικράτεια από την Πορτογαλία στο Αζερβαϊτζάν, γιατί μιλάμε για τέτοια έκθεση. Χρειαζόμαστε επίσης να εξασφαλίσουμε πως τα πανεπιστήμια έχουν πιο αποτελεσματική συνέχεια και παρακολούθηση του τι κάνουν οι απόφοιτοί τους. Και θέλουμε τη βοήθεια των Υπουργών σε αυτό. Να ξέρουμε κάθε στιγμή πού βρίσκεται ο απόφοιτος κάποιου πανεπιστημίου. Αυτό θα μας βελτιώσει στο να τους κάνουμε πιο απασχολήσιμους, δηλαδή να έχουν περισσότερες πιθανότητες να ε, μπουν στην αγορά. Και επίσης θα πρέπει να ζητήσουμε να ανοίξουν ε, το χώρο τους ανώτατης εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση με περισσότερε επαφέ με τον υπόλοιπο κόσμο. Κάθε δύο-τρία χρόνια συναντιόμαστε με υπουργό εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι αρκετό. Χρειαζόμαστε πιο τακτική συνεργασία, πιο πραγματικά μέτρα που θα ενισχύσουν τη συνεργασία και στο χώρο αυτό. Σα. ευχαριστώ πολύ κύριε Τάισεν. Θα δώσω τώρα το λόγο για πέντε λεπτά στο Λουίτζι αν το επιθυμεί. Εάν όχι, μπορούμε να κλείσουμε το θέμα. Λουίτζι. No, io, come diceva Cicerone, ho troppo abusato della vostra pazienza όπως ε, έχετε υπόψη σας, ε, μακρηγόρησα πριν, θα είμαι σύντομος τώρα. Εγώ έλαβα υπόψη μου το σύστημα της Γερμανίας. που λαμβάνει υπόψη την απασχολησιμότητα των ε, κατόχων πτυχίου bachelor από διάφορα πανεπιστήμια. Αν δείτε τα πτυχία bachelor και τη σχέση μεταξύ πανεπιστημίων και αγοράς εργασίας, μόνο 3% των πτυχιούχων bachelor δεν έχουν απασχόληση. Δεν το πίστευα, αλλά υπάρχουν στοιχεία Επίσης ε, διάβασα μια έκθεση της Ιταλικής Κονφιντούστρια με παρόμοια ευρήματα. Οπότε καταρχήν θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι γνωρίζουμε πολύ καλά την κατάσταση. Για την ηθαγένεια θα μιλήσω αργότερα γιατί καταλαβαίνω αυτό που μου είπατε. Αλλά ε, ε βέβαια θα καταθέσω τροπολογίες και θα πρέπει να βελτιωθεί η πρώτη πρόταση. Θα συνεργαστούμε για να συμφωνήσουμε όλοι επί ενό καλύτερου κειμένου. Ευχαριστώ πολύ. Η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών, είπα, είναι, είναι η 6η Δεκεμβρίου. Σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά ορισμένοι έχουν ήδη κάνει κάποιες σκέψεις και θα προλάβουμε. Και τον Ιανουάριο θα γίνει ψηφοφορία. Παρακαλώ και τον κύριο Μπερλιγκουέρ και τους συναδέλφους που θα καταθέσουν τροπολογίες να λάβουν υπόψη αυτά που είπε ο κύριο Τάισεν επίσης. Ότι δηλαδή θέλουμε ε, απτές και συγκεκριμένες προτάσεις εν ώψη του Βουκουρεστίου. Θα πρέπει να βάλουμε το δάχτυλο επί των τύπων των ύλων για να λειτουργήσει και να έχει αποτέλεσμα η Σύνοδο στο Βουκουρέστι. Κλείνουμε τη συζήτηση στο θέμα αυτό. Ξέρω ότι η κυρία Επίτροπος έχει ήδη έρθει. Ήρθε. Ανδρούλα, χαιρόμεθα διότι η Επίτροπος πριν πάει στο Συμβούλιο έρχεται σε εμά. Είμαστε και σημαντικότεροι κατά τη, τουλάχιστον σε αυτό το τομέα. Συζητήσαμε την uh, διαδικασία της Μπολόνια και την έκθεση του κυρίου Μπερλιγκουέρ και τώρα είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τις προτάσεις σας uh, του νέου προγράμματος uh, της, για τη διαβίου μάθηση. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Ντόρις, αγαπητοί φίλοι. Κυρίες και κύριοι, σήμερα θα σας παρουσιάσω μία πρόταση για ένα νέο πρόγραμμα εκπαιδευτικό το οποίο πέρασε ε, τις πρώτες συζητήσεις που κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ πάντα πίστευα πως ο ρόλος μου είναι να καταθέσω μία πρόταση η οποία θα είναι και συνεκτική και φιλόδοξη. Εάν η Ευρώπη αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει μία πιεστική ανάγκη να εκμετωρινήσει τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, να βελτιώσει τις δεξιότητες των λαών και να δώσει νέες ευκαιρίες στην νεολαία, τότε θα χρειαστεί αυτά να τα ε, φέρει στην επιφάνεια μέσω ενός προγράμματος που θα είναι άξιο των περιστάσεων. Αντί λοιπόν να έχουμε ένα μείγμα διαφορετικών δράσεων με διαφορετικό κύκλο ζωής του καθένα, θέλω να σας καταθέσω μία μακροπρόθεσμη στρατογική που θα έχει θετικές συνέχειες για χρόνια, για περισσότερες ευκαιρίες κινητικότητας, συνεργασίας και εταιρική σχέσης, με καινοτομίε για την χάραξη πολιτικής και με τη δημιουργία πολλών νέων εργαλείων που θα στηρίξουν τα κράτη-μέλη όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα ωφεληθούν από αυτές τις νέες ευκαιρίες. Ε, οποιοςδήποτε εργάζεται στο χώρο της λεωλέας, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, οι εκπαιδευόμενοι, ε, ε, όλοι οι φοιτητέ που στηρίζονται σήμερα, όλοι οι ενήλικες που είναι στη διαβίω εκπαίδευση, θα στηριχτούν περισσότερο από ό,τι σήμερα. Τι αλλάξαμε. Έχουμε ένα πρόγραμμα που είναι καλύτερο, κανόνες που απλουστεύθηκαν και βέβαια περισσότερους πόρους διαθέσιμου. Αυτό εγώ το θεωρώ πολύ καλό νέο. Νομίζω ότι θα ικανοποιήσει όλους. Και εδώ πρέπει να τονίσω το εξή: Κανείς από τους ενδιαφερόμενους δεν θα άντεται κάποια άλλη κατηγορία ενδιαφερομένων. Κανένας, όσο μεγάλος ή μικρός και να είναι, θα χρειαστεί να δώσει μάχη για να επιχορηγηθεί. Και νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό πλεονέκτημα που προσφέρει ένα ενιαίο πρόγραμμα όλοι αξίζουν προσοχής, όλοι αποτελούν τμήμα της κοινή προσπάθειας. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω μία ελάχιστη ε, πρικοδότηση για κάθε κατηγορία ενδιαφερομένων. Δηλαδή, δείτε το σε ένα ασφαλείας που εξασφαλίζει ότι σε κανένα κλάδο οι επιδοτήσεις δεν θα πέσουν κάτω από ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Στην πράξη δηλαδή, κάθε κατηγορία ενδιαφερομένων, κάθε ομάδα θα δει μία μεγάλη αύξηση στην καθαρή χρηματοδότηση που λαμβάνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα έχουμε ένα ενιαίο πρόγραμμα που θα μας επιτρέψει να αυξήσουμε την πρικοδότηση όλων. Δεν θα αφήσουμε κανέναν πίσω. Στην ανακοίνωση που συνοδεύει το νέο πρόγραμμα θα σας εξηγήσω πώς μπορούμε να κατανείμουμε τον προϋπολογισμό στις διάφορες ενδιαφερόμενες ομάδες. Θα ήθελα να τονίσω πως βεβαίως αυτά που σας περιγράφω τώρα είναι ενδεικτικά. Γιατί όσο τρέχει το πρόγραμμα βέβαια θα παρακολουθήσουμε και πώς οι διάφορες ομάδες χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα κονδύλια. Αυτή η προσωμείωση αποδεικνύει πως κάθε ενδιαφερόμενη ομάδα μπορεί να είναι και ε, νικηφόρα. Θα αυξήσουμε λοιπόν ε, την ε, χρηματοδότηση με τους εξής πολιτικούς στόχους. Στην ανώτατη εκπαίδευση που θα συμπεριλάβουμε και, τον, ε, και την επαγγελματική εκπαίδευση θα αυξήσουμε από το 85% στο 95% ε, την ε, τρέχουσα χρηματοδότηση. Άρα λοιπόν αποδεικνύουμε πως πιστεύουμε πως η ανώτατη εκπαίδευση θα προσφέρει και στην ανάπτυξη και στις θέσεις απασχόλησης και στην καινοτομία. Ε, για την διαβίου μάθηση και την επαγγελματική κατάρτιση θα αυξήσουμε 50 με 60% συγκρινόμενοι με την τρέχουσα χρηματοδότηση. Στα σχολεία θα αυξήσουμε 40 με 55% για την νεολαία. Εκτός από τις επιχορηγήσεις που λαμβάνουν από άλλους κλάδους, θα αυξήσουμε, μια, ε, θα αυξήσουμε μέχρι 40%. Και για την ε, διεθνή διάσταση της ανώτατης εκπαίδευσης θα φέρουμε μια αύξηση εκεί 17%. Όλα αυτά είναι δυνατά γιατί καταφέραμε να εξασφαλίσουμε η αύξηση του προπολογισμού μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βέβαια και χάρη στο ενιαίο πρόγραμμα που θα χρησιμοποιήσει κάθε ένα ευρώ για να εξυπηρετήσει μακροπρόθεσμους στόχους. Ένα ενιαίο πρόγραμμα ε, μας εξασφαλίζει μια απλούστευση στις προσπάθειες που κάνουμε έτσι ώστε όλοι οι Ευρωπαίοι να καταλαβαίνουν τι κάνουμε και να μπορούν εύκολα να ιτηθούν χρηματοδότηση. Το πρόγραμμα λοιπόν θα βασιστεί με τρία είδη δράσεων μόνο. Κινητικότητα για τη γνώση, συνεργασία και εταιρική σχέσεις και διάλογος για πολιτική. Αυτή η κινητικότητα για τη γνώση θα λάβει το μεγαλύτερο μερίδιο του συνολικού προϋπολογισμού, δηλαδή το 65%. Και είμαι πεπισμένη πως αυτή αποτελεί τη σωστή επιλογή, γιατί η κοινότητα η κινητικότητα είναι εκεί που η Ευρώπη μπορεί να φέρει την πραγματική διαφορά, τη μόνιμη διαφορά στις ανθρώπινες ζωές. Είναι ένα σημαντικό εργαλείο που θα εκμοντερνήσει τα ακαδημαϊκά ε, ιδρύματα σε όλα τα επίπεδα, σε όλη την Ευρώπη. Στο τέλος της τρέχουσας περίοδου, 400.000 άτομα θα έχουν χρησιμοποιήσει κατ' έτους τη δυνατότητα αυτή για κινητικότητα. Στο νέο προϋπολογισμό θα αυξήσουμε το επίπεδο αυτό σε ένα μέσο αριθμό 700.000 ατόμων το χρόνο για την επόμενη περίοδο του προϋπολογισμού. Και το 2020 ελπίζουμε και υπολογίζουμε πως ένα εκατομμύριο άτομα θα έχουν τη δυνατότητα τέτοιας κινητικότητας ε, στην Ευρώπη χάρη στις προσπάθειες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε να προτείνουμε και κάτι τελείω καινούριο μια, ένα μηχανισμό εγγυήσεων για τα φοιτητικά δάνεια που θα επιτρέπουν ε, σε περισσότερους μεταπτυχιακούς ε, φοιτητές να σπουδάζουν στο εξωτερικό. Γιατί αυτά τα μεταπτυχιακά βελτιώνουν τις δεξιότητες και ε, βοηθούν την καινοτομία. Μπορούν λοιπόν να παίξουν ζωτικό ρόλο στην ανάταξη των οικονομιών μας. Ας είμαστε σαφείς. Εμείς δεν θα προσφέρουμε αυτά τα δάνεια. Μαζί με την ΕΤΕ θα προσφέρουμε τις εγγυήσει για τα δάνεια που προσφέρουν οι επιλεγόμενοι ε, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί στα κράτη-μέλη υπό όρους βέβαια δανειακούς οι οποίοι είναι ε, πιο ευνοϊκοί από αυτούς που έχουν τα συνδυσμένα τραπεζικά δάνεια. Έτσι λοιπόν θα έχουμε ένα πολλαπλασιαστικό ε, αποτέλεσμα το οποίο θα είναι πιο αποδοτικό και λιγότερο ακριβό από τα παραδοσιακά δάνεια τα φοιτητικά. Δηλαδή θεωρούμε με ένα προϋπολογισμό 100 εκατομμυρίων το χρόνο θα επιτρέψουμε σε επιπλέον 55.000 φοιτητές μεταπτυχιακούς να σπουδάσουν στο εξωτερικό, να κάνουν το μεταπτυχιακό του στο εξωτερικό. Μετά την κινητικότητα, λοιπόν, το δεύτερο είδο δράσεων που θα στηρίξουμε είναι η συνεργασία και η εταιρική σχέση. Έχουμε σκοπό να στηρίξουμε ανάμεσα σε άλλε στρατηγικέ εταιρικέ σχέσει για μια μεγάλη γκάμα οργανισμών και φορέων που προσφέρουν κατάρτιση και εκπαίδευση και μεταξύ ε, ενώσεων νεολαία. Θα στηρίξουμε επίση μεγάλη κλίμακα ε, εταιρική σχέση μεταξύ τη εκπαίδευση και του επιχειρηματικού κλάδου. Θα είναι συμμαχίε υπέρ της ε, για την ανώτατη εκπαίδευση, την ανώτερη εκπαίδευση και για δεξιότητε που χρειάζονται διάφοροι βιομηχανικοί κλάδοι και θα ε, προωθήσουμε την ηλεκτρονική αδελφοποίηση όπως επίσης και ε, πλατφόρμες υψηλής τεχνολογίας. Δηλαδή, δημιουργία δυναμικού σε τρίτες χώρες, αυτό επίσης θα στρίριχθει, εστιάζοντας κυρίως στη δική μας ευρωπαϊκή γειτονιά. Να το εξηγήσω. Εταιρική σχέση μεταξύ ε, βιομηχανίας και ανώτατων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Έτσι λοιπόν θα έχουμε νέους τρόπους παραγωγής ε, και κατανομής της γνώσης, δημιουργικότητα, επτερικό ε, και ε, επιχειρηματικό πνεύμα, νέα πανεπιστημιακή ύλη και νέα προσόντα. Θέλουμε να εστιάσουμε επίσης την προσοχή μας και να προωθήσουμε την ευρωπαϊκή διάσταση στα σχέδια εθελοντισμού στα διάφορα κράτη-μέλη. Και εδώ χρειάζεται η διεθνής κινητικότητα. Θέλουμε εταιρική σχέση μεταξύ περιφερειακών και τοπικών αρχών, έτσι ώστε να εμπλακούν παίκτες και ομάδες από διάφορους κλάδους και να προωθήσουμε νέες στρατηγικές για τη διαβίου μάθηση, πιο αποτελεσματική χρήση των πόρων και κάποια καθεστώτα κινητικότητα τα οποία θα είναι πιο ποιοτικά. Και αυτή είναι αυτό είναι ένα μικρό αριθμό των εταιρικών σχέσεων που έχουμε κατά νου. Γιατί βεβαίω έχουμε και τον διάλογο σε επίπεδο πολιτικής πέραν της κινητικότητας και της συνεργασίας. Εδώ θα μοιράσουμε ε, και κείμενα όπου θα έχουμε τις βέλτιστες πρακτικές και τις νέες ιδέες. Για να πετύχουμε τους μακροπρόθεσμους στόχους στην παιδεία και στην κατάρτιση, χρειαζόμαστε οι πολιτικές μας να είναι ευφυείς, να αναλύουμε τι συμβαίνει σε κάθε χώρα και να έχουμε ένα είδος ε, πολυμερούς παρακολούθησης. Πρέπει να διδαχθούμε από κάθε ευρωπαϊκή χώρα και αυτό όταν έχει γίνει στο παρελθόν έχει ε, προωθήσει την ποιότητα των επενδύσεών μα και έχει παροτρύνει τα κράτη-μέλη να σχεδιάσουν καινοτόμε πολιτικέ. Προτείνω λοιπόν να ε, στοχεύσουμε σε μία σειρά προτεραιοτήτων σε όλου του κλάδου. Δηλαδή, μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνουμε τον ε, εξυγχρονισμό της ανώτατη εκπαίδευση, τη διαδικασία τη Μπολόνια, τα βασικά προσόντα που προσφέρει η διαβίου μάθηση, ε, το νέο βαθμολογικό πίνακα για τα πανεπιστήμια, την υψηλή τεχνολογία στα σχολεία, ε, να προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα που έχει η εγκατάλειψη, η του σχολείου σε μικρή ηλικία, επίσης να προωθήσουμε την γνώση ξένων ε, γλωσσών και να έχουμε ε, καλύτερες επιδόσεις στον αλφαβητισμό. Θα πρέπει λοιπόν αυτή την θέση της Ευρώπης, την προωθημένη, να την εντάξουμε στην εξωτερική διάσταση του προγράμματός μας. Μεγαλύτερη συνεργασία με τρίτες χώρες. Να ευθυγραμμίσουμε τη δουλειά που κάνουμε τις τρεις βασικές κομβικές δράσεις του νέου προγράμματος με πολύ μεγάλη έμφαση που θα δοθεί στην κοινοτικότητα. Να πούμε πως αυτά τα κοινά πτυχία που στηρίζουμε σε όλο τον κόσμο θα διευρυνθούν και θα γίνουν πολλά περισσότερα. Θεματικές και ογραφικές προτεραιότητες στα πλαίσια της εξωτερικής μας πολιτικής. Διανύουμε το χρόνο της αραβικής Άνοιξης. Και χαίρομαι που θα ανακοινώσουμε μια ενισχυμένη συνεργασία με χώρες ε, όμορες ε, στο Νότο και στην Ανατολή. Θα στηρίξουμε την ε, αύξηση του δυναμικού των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εκεί και τον εξυγχρονισμό της ανώτατης παιδείας και θα σχετίσουμε αυτές τις δράσεις με την, με την κινητικότητα και του προσωπικού των ιδρυμάτων αυτών, αλλά και των φοιτητών. Θέλω να πω και δύο λόγια για την νεολαία και τον αθλητισμό. Θα ολοκληρώσουμε τις βασικές μας δράσεις στη νεολαία με το νέο πρόγραμμα, χτίζοντας γέφυρες μεταξύ της άτυπης γνώσης και της ε, ε απόκτησης ε, ε, προσόντων μέσω της ανταλλαγής νέων, μέσω του ευρωπαϊκού διθελοντισμού και, του, και της υπηρεσίας μέσω της διαδικτύωση και δικτύωση των νέων και θα συνεχίσουμε με το διαστρωμένο διάλογο που έχουμε ξεκινήσει με τι ενώσει νεολαίας. Ελπίζω αυτό να ήταν σαφέ. Δεν θέλουμε να υποσκάψουμε την δουλειά που κάνουν οι ομάδε νέων ε, στην συμμετοχή και στην εκμάθηση και εξοικείωση με τη δημοκρατία. Αντίθετα, στηρίζουμε τι προσπάθειε του, διευρύνουμε του πόρου και δίνουμε περισσότερε ευκαιρίες. Ο αθλητισμό για πρώτη φορά αποκτά το δικό του κεφάλαιο και δικό του προπολογισμό και θα κάνουμε πολλές και διαφορετικές δράσεις. Προτείνουμε εδώ ένα μέσο ετήσιο προϋπολογισμό 30 εκατομμυρίων ευρώ. Έτσι θα μπορέσουμε να στοχεύσουμε σε θέματα τα οποία δεν μπορούν με αποτελεσματικό τρόπο να λυθούν στο ε, εθνικό επίπεδο. Το πρόγραμμα θα καλύψει στόχους που έχουν μεγάλη ε, κοινωνική και οικονομική επίπτωση. Ε, καλή διακυβέρνηση, ε, πλεονεκτήματα και ωφέλη για την υγεία, κοινωνική ένταξη, διπλές προοπτικές καριέρας για τους αθλητές και βέβαια οι διεθνείς απειλές του ντόπινγκ, των στημένων, της βίας και του ρατσισμού και για το όνομα του προγράμματος θέλαμε να φάνε κάτι το οποίο θα είναι αναγνωρίσιμο. Όχι μόνο στις Βρυξέλλες, όχι μόνο ε, στο δικό μας ε, κοινό, αλλά αναγνωρίσιμο και από τον πληθυσμό, ε, από τους λαούς της Ευρώπης. Θέλαμε κάτι το εμβληματικό, που θα συμβολίζει τις ε, καλύτερες επιτυχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, κάποια σήμα που θα θέλουν και οι υπόλοιποι να δανειστούν. Θέλαμε όμως να ε, υπογραμμίσουμε τις νέες ευκαιρίες που όλοι θα έχουν στη διάθεσή τους. Οι ενδιαφερόμενοι στην παιδεία, στην κατάρτιση, στην νεολαία, στον αθλητισμό και γι' αυτό το νέο πρόγραμμα θα το πούμε «Εράσμους για όλους». Erasmus for All στα αγγλικά. Τον Ιούνιο φέτος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ο προϋπολογισμός ο δικός μας να αυξηθεί ε, κατά 73% περίπου. Μεταξύ του 2014 και του 2020 προτείνουμε να επενδύσουμε παραπάνω από 17 δις ευρώ στο μέλλον των λαών μας το ποσό αυτό είναι υψηλότερο ακόμα και αυτό το οποίο ανακοινώσαμε τον Ιούνιο. Γιατί έχει ε, προσαρμοστεί ε, στον πληθωρισμό και έχει συμπεριλάβει και τη διεθνή διάσταση. Ο νέος αυτός προϋπολογισμός φέρνει μια αλλαγή χωρίς προηγούμενο στις πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι μια αλλαγή την οποία όλοι πρέπει να χαιρετήσουμε, γιατί τη στιγμή που η Ευρώπη αντιμετωπίζει μία από τις βαθύτερες και πιο ανησυχητικές κρίσεις, είναι καθήκον μας να προτείνουμε ελπίδα για το μέλλον. Δεν μπορώ να φανταστώ από ε, καλύτερο, τρόπο από επενδύσεις στην παιδεία, στην κατάρτιση που θα προσφέρει σε όλους, σε όλες τις ηλικίε από οπουδήποτε και αν προέρχονται, τη δυνατότητα ε, να ε, χρησιμοποιήσουν τις ευκαιρίες που τους προσφέρουμε και να παίξουν τον πλήρη ρόλο που τους ανήκει στην κοινωνία. Για όσους επιχειρηματολόγουν και λένε πως ξεχνάμε ποιο είναι ο κοινωνικός ρόλος της εκπαίδευσης, την εκπαίδευση για τη γνώση, θα τους ρωτήσω, έχει άραγε κοινωνικό ρόλο ρόλο αυτή η ανεργία στους νέους που έχει φτάσει στο 40%. Γιατί η ανθρώπινη κρίση που αντιμετωπίζουμε σε κάποιες χώρες. Είναι μια αποστολή την οποία με κάποιο τρόπο πρέπει να αναλάβουμε. Ε, αυτή η αύξηση του 73% μην νομίζετε, μην νομίζετε πως μας προσφέρθηκε εύκολα και ανοιχτόχερα. Χρειαστήκαμε να σχεδιάσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα μεγιστοποιήσει την επίπτωση κάθε ευρώ που θα δαπανηθεί. Πολύ συχνά στο παρελθόν ανακοινώσαμε ότι είναι πολύ σημαντική η νεολαία, η ε, εκπαίδευση, η κατάρτιση και μετά δεν χρηματοδοτήσαμε επαρκώς. Σήμερα τα πράγματα άλλαξαν. Σας φέρνω μια πρόταση που προσφέρει τεράστιες ε, ευκαιρίες σε κάποιες από τις πιο κομβικές ε, κάποια από τα πιο κομβικά κοινωνικά ε, ιδρύματα και σε εκατομμύρια ανθρώπους που ανησυχούν για το ποιο θα είναι το μέλλον τους. Σήμερα λοιπόν θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει ε, με αυτό το οποίο σας προτείνουμε. Μία χωρίς προηγούμενο αύξηση ε, προϋπολογισμού για όλους τους ενδιαφερόμενους, μία τολμηρή, ένα τολμηρό πρόγραμμα που θα ανταποκριθεί στι ανάγκες Ελπίζω στις δύσκολες συζητήσεις που θα γίνουν στο μέλλον να μας βοηθήσετε. Για κάθε πρόταση σίγουρα δεν θα συμφωνήσουμε, αλλά πιστεύω ειλικρινά πως οι στόχοι που μοιραζόμαστε μας ξεπερνούν, ε, ξεπερνούν τις διαφορές μας. Ε, θα ήθελα τώρα να πω και δύο λόγια, αγαπητοί φίλοι, για ένα νέο πρόγραμμα στον πολιτισμό που λέγεται «Η Δημιουργική Ευρώπη», Creative Europe. Ελπίζω, νομίζω ότι θα με καταλάβετε που δεν θα σας πω τόσα όσα είπα για την εκπαίδευση, γιατί εδώ δεν προτείνουμε κάτι το τόσο καινοτόμο και οι προηγούμενες συζητήσεις που κάναμε απέδειξαν ότι υπάρχει ευρύτερη συνένεση για τα κύρια σημεία του προγράμματος. Θα σας προτείνω σήμερα ένα πρόγραμμα το οποίο διατηρεί την εμβληματική ταυτότητα των δύο τμήματων, τα ΜΜΕ και ο πολιτισμός θέλουμε μία υπηρεσία ενιαίας εξυπηρέτησης για όλες τις πολιτιστικές και δημιουργικές δραστηριότητες με διαφορετικές πύλες εισόδου για τον πολιτισμό και τα μίντια ε, που φασίζεται στις δικές τους ανάγκες. Έχουμε όμως και μία τρίτη πύλη που θέλει να βοηθήσει τους, ε, δημιουργικές, ε, τους δημιουργικούς κλάδους μας. Το νέο αυτό μέσο θα αυξήσει τον αριθμό των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που γνωρίζουν τα θέματα και ε, στους χώρους του πολιτισμού και της τέχνης ε, να τα διευρύνει σε γεωγραφικό επίπεδο και να μοχλεύσει τις ιδιωτικές επενδύσεις που κάνουν. Επίσης θέλουμε να αλλάξουμε το συμπερι... τη συμπεριφορά κάποιου ε, τμήματος ε, της σχετικής, των σχετικών κλάδων στην Ευρώπη, να τους απομακρύνουμε από τις επιχορηγήσεις και να τους πρόξουμε προς, τα δάνεια. The objectives of Creative Europe are Θέλουμε να στηρίξουμε την ε, ικανότητα των πολιτιστικών και δημιουργικών ε, βιομηχανιών να λειτουργούν σε διεθνές επίπεδο, να προωθήσουμε την διασυνοριακή κυκλοφορία πολιτιστικών και δημιουργικών έργων να βοηθήσουμε τις ε, επιχειρήσεις ε, αυτές να και τις εταιρείες να αποκτήσουν νέα κροατήρια στην Ευρώπη και εκτός Ευρώπης, να ενισχύσουμε την οικονομική ικανότητα των τομέων της δημιουργικότητας και του πολιτισμού, να ενισχύσουμε την πολιτική συνεργασία. Ο τομέας του πολιτισμού θα συνεχίσει να στηρίζει προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας. Για την περίοδο 2014-2020, τουλάχιστον 8.000 πολιτιστικές οργανώσεις, οργανισμοί θα συμμετάσχουν σε προγράμματα συνεργασίας. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι οι μικροί πολιτιστικοί οργανισμοί θα είναι εξίσου ευπρόσδεκτοι όπως όλοι οι άλλοι. Σε ό,τι αφορά τώρα ε, για τα μέντια. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τη διανομή ευρωπαϊκών ταινιών, κινηματογραφικών ταινιών. Θα βοηθήσουμε τον τομέα να ε, υποστηριχθεί και να ωφεληθεί από την ψηφιοποίηση και θα ανοίξουμε σε νέους τομείς όπως video games. Ε, ενσωματώνοντας το πρόγραμμα Media Mundo, το κομμάτι Media θα ενθαρρύνει ε, οι επαγγελματίες στον οπτικοακουστικό τομέα να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους και εκτός Ευρώπης. Κυρίες και κύριοι, η Κομισιόν προτείνει σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού για αυτό το πρόγραμμα το καινούριο. Ένα ε, συνολικό ποσό 1,8 δις ευρώ που σημαίνει 37% αύξηση στις τρέχουσες δαπάνες. Η αύξηση αυτή ε, είναι μια σαφής απόκριση προς τις προτεραιότητες της στρατηγικής ε, Ευρώπη 2020. Επενδύοντας στις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες μας, συμβάλλουμε απευθείας ε, στις προσπάθειες προς την έξυπνη, βιώσιμη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Το 2008 οι τομεί δημιουργική και πολιτιστική ήταν το 4,5% του ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και απασχολούσε περίπου το 4% του ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού. Οι κλάδοι αυτή είναι επίση ζωτική σημασία γιατί ε, φέρουν ωφέλη και σε άλλου τομεί διότι δίνουν περιεχόμενο για τις νέες τεχνολογίες, συνδυάζουν και συμβιβάζουν την κοινωνική ένταξη και τη διαφορετικότητα και ε, προωθούν την κοινωνική καινοτομία. Αν όμως θέλουμε να αξιοποιήσουν το δυναμικό τους για περαιτέρω ανάπτυξη, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βοηθήσει να δημιουργηθούν οι σωστέ συνθήκες προϋποθέσεις. Και αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε με την δημιουργική Ευρώπη Creative Europe και ελπίζω ότι θα δώσετε την πλήρη υποστήριξή σα στο καινούριο πρόγραμμα. Ευχαριστώ αγαπητή Ντόρι, ευχαριστώ αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι. Ε, αυτή είναι, αυτό είναι ένα ε, χειροκρότημα για την καλή δουλειά που κάνετε, την ωραία παρουσίαση, όχι όμως 100% ε, για το περιεχόμενο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Στούβια. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ την Επίτροπο και αυτή την έκθεση που μας έκανε εδώ. Αυτό των νέων προγραμμάτων μας παρουσίασε θα προσπαθήσω να είμαι αρκετά σύντομος, γιατί υποθέτω πολύ θέλω να παρέμβω από συναδέλφους και θα προσπαθήσω να είμαι πραγματικά λακωνικός για τα θέματα που θέλω να εξετάσω. Ας αρχίσουμε αυτά που μου αρέσουν. Είμαι πάρα πολύ ευτυχής ότι υπάρχει μια αύξηση αυτή τη στιγμή του προπολογισμού και αυτό είναι ένα σημάδι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί φαίνεται ότι θέλουμε να απαιτήσουμε στους νέους, στην κουλτούρα, στον πολιτισμό, στην ε, ε, ε. Επίσης μου ικανοποιεί το γεγονός ότι έχει εισαχθεί η προσπάθεια η οποία έχει γίνει και νομίζω πως πραγματικά εμείς στο Κοινοβούλιο και η Κομισιό που έχει επιμείνει σε αυτό το σημείο έχει συμπεριληφθεί μέσα στην έκθεση. Επίσης οι στόχοι, γενικότεροι στόχοι μου ικανοποιούν πάρα πολύ. Διότι κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να φτάσουμε καλύτερα στους στόχους στους οποίους έχουμε προκαθορίσει σε αυτά τα προγράμματα. Πρέπει να σας πω ακόμη, αυτό που δεν μου αρέσει τόσο είναι αυτή, είναι ο ένας προγραμματισμός αυτός, ωστόσο η εξαφάνιση των ονομα, μερικών ονομάτων για το πρόγραμμα στις, για τους νέους ε, το Εράσμος είναι ένα, μια, ένα σήμα ιστορικό, το ξέρουμε όλοι, έχει, έχει αποδειχθεί και λειτουργεί βεβαίως και αυτό το καινούριο για το learning είναι όλα αυτά σύμβολα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σήμερα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες για αυτή τη το, Αυτή η έλλειψη όμως συντονισμού μεταξύ όλων αυτών μπορεί να δημιουργήσει μια σύγχυση καθότι οι νέοι τουλάχιστον σε αυτό το σχήμα το οποίο παρουσιάστηκε εδώ το πρόγραμμα ότι οι φοιτητέ μπορούν να να μπουν όλοι φοιτητέ, ερευνητέ, μεταπτυχιακοί κλπ. σε αυτό το πρόγραμμα. Νομίζω ότι πραγματικά είναι κάτι το οποίο δεν είναι σωστό και μας διαφεύγει η προσπάθεια που θα πρέπει να γίνει και θα έπρεπε να είναι πιο συστηματική. Νομίζω πως θα πρέπει να υπάρξει ένα πρόγραμμα για τους νέους και μόνο, και γιατί αυτό είναι κάτι σημαντικό. Δεν υπάρχουν βέβαια όλα τα σημεία εκείνα που πρέπει να υπάρχουν και υπάρχουν δύο περιβάλλοντα τα οποία, δύο πτυχές αν θέλετε, οι οποίες είναι διαφορετικές και οι στόχοι μεταξύ των μεν και το δε είναι διαφορετικές, εκεί που αποβλέπουν είναι κάτι το διαφορετικό, νομίζω πως πραγματικά οι καθηγητές, οι ερευνητές, οι νέοι, δεν νομίζω πως πραγματικά μπορούμε να τους βάλουμε όλους αυτούς στον ίδιο κόρβανα δεν είναι από τις βέλτιστες ιδέες που υπάρχουν μέσα στην έκθεση. Επίσης θα ήθελα να υπογραμμίσω και κάτι ακόμη όσον αφορά την, αυτή τη δημοσίευση που γίνεται για συμπληρωματικό δρόμο, διότι υπάρχουν ε, για αυτές τις διοικητικέ απλοποιήσεις που θέλουν να γίνουν και βεβαίως με αυτές τις ε, οργανώσεις των νέων, αυτές τις εταιρισμού των νέων και νομίζω πραγματικά μερικές φορές είναι πάρα πολύ δύσκολο να τους βάλουμε όλους αυτούς, να τους συμπεριλάβουμε μέσα σε ένα κεφάλαιο. Αυτό το project λοιπόν νομίζω απομακρύνει όλο και περισσότερο αυτοί, αυτούς οι οποίοι θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα, τους αποξενώνει αν θέλετε. Έτσι λοιπόν αυτή η τεχνική πρόταση η οποία γίνεται στο κεφάλαιο αυτό που έχει βλέπουμε ότι πραγματικά προπολογισμό είναι ένα, ένα δις 800 εκατομμύρια νομίζω πως πραγματικά μπορούμε να δούμε εάν κάνουμε το σύνολο λείπει κάτι λείπει κάτι και δεν ξέρω πραγματικά τι είναι αυτό το ποσό το, το οποίο μπορεί να έχει ε, δει πάει αλλού για να συμπεράνω κύριε Επίτροπε. Έχω πολλά να πω βεβαίω, αλλά υπάρχουν πολλά πράγματα που είναι καλά, υπάρχουν μερικά όμως όπως σας είπα τα οποία είναι λιγότερο καλά θα τα χαρακτηρίζα. Δεν μου αρέσει το όνομα ερά, το Εράσμους, αυτό το γενικό Εράσμους που διαγράφει όλα τα ονόματα τα προηγούμενα και τα σήματα που υπήρχαν και μπορούν να δημιουργήσουν, μπορεί να δημιουργήσει αυτό περισσότερη σύγχυση μεταξύ των φοιτητών ή των ενδιαφερόμενων που θέλουν να συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Καμέιβα. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζω μετά τον προηγούμενο ομιλητή γιατί έχω παρόμοια προβλήματα Πρώτα όμως πρέπει να πω ότι μας έχετε όλους στο πλευρό σας ε, όταν δίνετε μάχες για αύξηση του προϋπολογισμού ε, και θέλετε να τις επιβάλλετε στο Συμβούλιο Υπουργών που θα είναι σκληρός αγώνας. Σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση των προγραμμάτων ε, υπάρχουν ανοιχτά ερωτήματα και προβλήματα σε σχέση με τις προτάσεις σας. Ε, εράσμους για όλους. Και εμένα δεν με πείθει γιατί το Εράσμους είναι πια ένα σύμβολο, ένας, μια γνωστή έννοια στην Ευρώπη που αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση, πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Στο Erasmus for All συμπεριλαμβάνομαι όλη την εκπαίδευση. Οπότε θα δημιουργηθεί και η λάθος εντύπωση στην Ευρώπη ότι πρόκειται μόνο για την πανεπιστημιακή ή τριτοβάθμια εκπαίδευση και εδώ. Οπότε αυτό δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει. Πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε διακρίσεις. Επίσης, ελάχιστες ε, ε, πρικοδοτήσεις για κάθε τομέα. Πώς δηλαδή θα είναι αυτές οι ελάχιστες ε, ε, ε, κατανομές των κονδυλίων, των πιστώσεων και πώς θα γίνει αυτό από την άποψη της τεχνικής κατάρτισης του προϋπολογισμού στις επιμέρους γραμμές θα συνεχίσουμε να έχουμε επιμέρους γραμμές του προϋπολογισμού και ποιος θα αποφασίζει για τα χρήματα τα οποία υπερβαίνουν τις ελάχιστες αυτές πιστώσεις, ε, αυτά που θα περισσεύουν. Εμείς θα θα κάθε χρόνο με αυτό το θέμα ως κοινοβούλιο ή θα το αναθέσουμε στην Κομισιόν, ε, κάτι που νομίζω ότι δεν το θέλει κανείς μας. Δηλαδή, πώς θα γίνει δημοσιονομικά αυτή η διαδικασία, η άσκηση αυτή. Είναι ενδιαφέρον αυτό, γιατί μα ενδιαφέρει ω Κοινοβούλιο να μπορούμε να αποφασίζουμε κι εμείς πόσα χρήματα θα διατίθενται για ποιε γραμμές προγραμμάτων, έργων, projects και πού θα δίνονται οι προτεραιότητες. Και όλα αυτά με τρόπο ε, ε, που να ε, διευκολύνει την εποπτεία. Επίσης, δεν θα υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ μικρών και μεγάλων εντάξει, θεωρητικά ως δήλωση ωραία, ωραία ακούγεται, αλλά στην πράξη δεν το πολύ πιστεύω, γιατί όταν όλα τα προγράμματα που είχαμε μέχρι τώρα ε, ειδωθούν από κοινού, τότε τα προγράμματα για την νεολαία δεν θα ανταγωνίζονται με μεγάλα πανεπιστήμια, ας πούμε, που ε, έχουν συνεργασία για ερευνητικά προγράμματα. Υπάρχει μεγάλη έλλειψη ισορροπίας σε ό,τι αφορά τους ετούντες. Άρα λοιπόν τα μικρότερα projects που θα έχουν μικρότερες πιστώσεις, λιγότερο ε, προσωπικό, δεν θα μπορούν να είναι ανταγωνιστικά. Και προφανώς αυτό είναι κάτι που δεν το θέλουμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Λότεγκαρτ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Καταρχήν συγχαρητήρια η πρόταση και το πρόγραμμά σας είναι η πιο φιλόδοξη προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η τωρινή κρίση. Είναι ένα σημαντικό και εντυπωσιακό βήμα μπροστά και νομίζω ότι Πράγματι πρέπει να κάνει κανείς προσπάθεια για να είναι απεσιόδοξος εδώ. Βλέπω ότι είναι κάποιοι, αλλά τα δείγματα γραφής είναι καλά και νομίζω ότι θετικά πρέπει να κρίνουμε το αποτέλεσμα μέχρι τώρα. Επίσης πιστεύω ότι φαίνεται οι προτεραιότητες που θέσατε να είναι οι σωστές Σωστό είναι να βελτιωθεί το κομμάτι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και το 65% κινητικότητα είναι επίσης σωστό ποσοστό και στηρίζουμε ως ομάδα την προσπάθειά σας να εξυγχρονίσετε την κατάσταση. Είναι πολύ καλό να υπάρχει ένα όνομα για το πρόγραμμα αυτό. Τώρα, θα επιστήσω την προσοχή σας σε έναν άλλον τομέα που μας απασχολεί ξέρω ότι το ξέρετε εσείς, δεν ξέρω αν το ξέρουν οι συνάδελφοι, αλλά όλη η ιδέα της εστίασης στις εξωτερικές σχέσεις είναι επίσης πολύ καλή. Και έχω μία ερώτηση σχετικά. Φαίνεται, αν δούμε την Κίνα για παράδειγμα, φαίνεται ότι η Επιτροπή Πολιτισμού ε, έχει να συμβάλλει στις σχέσεις ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά είναι ο τρίτος πυλώνα στην Κίνα η ε, εκπαίδευση, κατάρτιση και θα πρέπει να την εξετάσουμε τη χώρα αυτή για να δούμε πώς θα βελτιώσουμε τις σχέσεις με τη χώρα και να να αντιμετωπίσουμε και την κρίση. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα της εκπαίδευσης ε, στο πυλώνα. Έχουμε τώρα τη δυναμική για να το κάνουμε αυτό και νομίζω ότι το παρόν πρόγραμμα είναι το σωστό μέσον. Επίσης, ε, επίκειται και ο διαπολιτιστικός διάλογος ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας Οπότε είναι η ευκαιρία να το κοιτάξουμε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό ο ρόλος του πολιτισμού για να βγούμε από την κρίση και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την Κίνα ως μέσον. Ε, πήγα πρόσφατα στη Σανγκάη και επισκέφθηκα το Πανεπιστήμιο Φουτάν και το την επιχειρηματική σχολή Κίνα, Συνοευρωπαϊκή. Ε, πολύ σημαντικά πανεπιστημιακά ιδρύματα και είδα από τις συνομιλίες μου ότι είναι διατεθειμένοι να ενισχύσουν τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το πρόγραμμα λοιπόν και τα αυξημένα κονδύλια για το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθούν πολύ αποτελεσματικά και εδώ. Να πάω στην ερώτησή μου τώρα. Κοιτάζοντας τα νούμερα, βλέπω 17% αύξηση της ε, διεθνούς διάστασης. Και αναρωτιέμαι, Βλέποντας τα νούμερα, βλέπω ότι 200 μόνοι ε, φοιτητές από την Ευρωπαϊκή Ένωση πήγαν στην Κίνα φέτος. Είναι πάρα πολύ χαμηλός ο αριθμός αυτός. Μπορούμε να τον αυξήσουμε κατά πολύ. Ερωτώ λοιπόν, αυτό σας απασχόλησε όταν ε, δουλεύατε στο το πρόγραμμα και έχετε συγκεκριμένα προγράμματα για τη βελτίωση και ενδυνάμωση αυτής της συνεργασίας, γιατί έχουμε κάποιες εξαιρετικές ευκαιρίες για να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας με την Κίνα σε αυτό το τομέα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριος Φίσες. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, και θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Επίτροπο. Θα ήθελα να συνταχθώ με τα όσα είπαν οι προλαλήσαντες συνάδελφοι. Καταρχήν θα ήθελα να σας συγχαρώ. Να σας συγχαρώ για την αύξηση αυτή του προπολογισμού σε μια στιγμή κρίσης. Νομίζω για σας είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Και είμαι σίγουρος πως ήταν πολύ δύσκολο πραγματικά αυτή την αύξηση ε, να την ε, πετύχετε ε, που τους υπολείπους συναδέλφους σας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το θέμα το οποίο εμένα με ανησυχεί είναι κάποια προγράμματα τα οποία θα καταργηθούν. Νομίζω το να έχει κανείς κάποιο εμπορικό σήμα για να χαρακτηρίσω έτσι την ονομασία κάποιων προγραμμάτων είναι μια προσπάθεια που κάνουν όλες οι εμπορικές εταιρείες ε, και το να καταργήσουμε εμείς κάποια προγράμματα ε, θα δημιουργήσει σύγχυση. Δηλαδή να το πω διαφορετικά. Για το πρόγραμμα που επιλέξατε, ίσως θα έπρεπε να το ονομάσετε διαφορετικά για να μην δημιουργήσει πρόβλημα με το προηγούμενο Εράσμους. Γιατί το Εράσμους Μούντους ή το Κομένιους, το Λεωνάρδος, το Lifelong Learning Εράσμους είναι πολύ γνωστά. Όλοι ξέρουν ποια είναι τα προγράμματα αυτά. Και για μένα είναι σφάλμα να εξαφανιστούν αυτές οι ονομασίες γιατί αν δεν έχουν ε, συγκεκριμένο φάκελο και πρικοδότηση για το Erasmus Mundus και το Erasmus το απλό και το Erasmus Lifelong Learning, όλοι τα ξέρουν παντού, όλοι οι φοιτητέ. Όλοι έχουν κάνει έρασμο και νομίζω ότι θα δημιουργήσει σύγχυση ε, γιατί είναι πολύ πετυχημένα. Μην τους δώσετε λοιπόν αυτή την γενικότερη ονομασία που θα συμπεριλαμβάνει το όνομα Erasmus Και για τα όσα είπε ο συνάδελφος, το Marie Curie λείπει. Και αυτό δεν είναι σημαντικό για την επιστημονική έρευνα. Δεν θέλω να μακρηγορήσω. Σας συγχαίρω πάντως. Σας συγχαίρω και για τον αθλητισμό. Για πρώτη φορά, όπως είπατε και εσείς, έχουμε ε, έναν ικανό προϋπολογισμό και πιστεύω πως ε, εδώ το πιο βασικό είναι ότι καταφέρατε ο αθλητισμός να θεωρηθεί ε, πως είναι ισότιμο σκέλος των υπόλοιπων που έχετε στο πρόγραμμα. Γιατί στον αθλητισμό κυκλοφορούν πολλά χρήματα. Βέβαια τα κράτη-μέλη θα αποφασίσουν πώς θα χρησιμοποιήσουν την πυργοδότηση που θα τους δώσετε είτε για τον αθλητισμό είτε για κάποια άλλη πτυχή. Αλλά και η απλή συμπερίληψη του αθλητισμού στα ταμεία αυτά είναι μία νίκη. Ευχαριστώ κύριε Μπόρις. Αξιότιμη κυρία Επίτροπε, θέλω να σας συγχαρώ θερμά. Ήταν αυτή μια ανέλπιστη επιτυχία για μας εν ώψη της γενικευμένης κρίσης. Οι νέες ονομασίες ε, για τα δύο προγράμματα ε, ε, λυρώνουν αυτό που περιέχει η στρατηγική για την Ευρώπη του 2020. Θα ήθελα να μου πείτε το εξής. Ορισμένα προγράμματα όπως το Marie Curie δεν βρήκαν θέση. Εμείς λαμβάνουμε πολλά σήματα και μηνύματα από νέους που ανησυχούν γιατί δεν γνωρίζουν αν, για παράδειγμα, το, το πρόγραμμα Media θα ε, συνεχίσει να διατηρεί μια κάποια ανεξαρτησία που είχε. Θα ήθελα λοιπόν μια συγκεκριμένη πληροφορία για τη συνέχιση που θα δώσετε, ε, στη συνέχεια που θα δώσετε στο πρόγραμμα αυτό. Επίσης, ε, δεν έχουμε πληροφορίες για τα διαρθρωτικά ταμεία. Όμως θα θέλαμε να πούμε το εξής. 6 δις ευρώ ήταν τα κονδύλια που χρησιμοποιήσαμε από τα διαρθρωτικά ταμεία για τον πολιτισμό. Στο κανονισμό για τη νέα δημοσιονομική περίοδο παρατηρούμε ότι δεν μπορούμε πια να επενδύουμε στον κινηματογράφο σε άλλα πολιτιστικά αγαθά. Από το παρουσιάσατε τις δαπάνες από το, σύλλογο, από σύνολο του προϋπολογισμού, αλλά υπάρχουν μειώσεις και περιορισμοί στα πλαίσια των διαρθρωτικών ταμείων. Ε, ευχαριστώ. Η κυρία Μανέσκου, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε κυρία Επίτροπε. Ευχαριστώ την Επίτροπο για την ομιλία της και την συγχαίρω για το πρόγραμμα που είναι μεγάλο βήμα μπροστά για την διασφάλιση του μέλλοντος του πολιτισμού στην Ευρώπη, ιδιαίτερα τώρα με την κρίση. Χαιρετίζω το νέο πλαίσιο των προγραμμάτων, διότι επιτρέπει περισσότερες επενδύσεις αναφέρατε το 73%. Επίσης ε, μιλήσατε και για τα παιδιά που εγκαταλείπουν το σχολείο, για τη βελτίωση επίσης της εκπαίδευσης στα σχολεία και πρέπει να συνεχίσουμε να επενδύουμε γενικότερα για την υποστήριξη των νέων μέσα από διάφορες δράσεις, γιατί είναι η πιο ευάλωτη κατηγορία που, έχει, που πιο πολύ από άλλες από την κρίση. Υπάρχουν και εθνικά προγράμματα, υπάρχουν ε, κινήματα των νέων που μπορεί να προωθηθούν μέσα από το ευρύτερο αυτό πλαίσιο ε, δεν ξέρω αν μπορούμε να αναδεικνύουμε επιμέρους τομείς, όπως για παράδειγμα ε, την όλη προβληματική του Youth in Motion, ε, η συγκίνηση. Και επίσης οι μικρές ενώσεις και οργανώσεις νέων που έχουν μικρά προγράμματα θα, δεν θα ωφεληθούν. Γιατί αυτοί όμως αποτελούν ένα μεγάλο κομμάτι του ε, Youth in Motion. Επίσης, ε, οι νέοι από ευάλωτα κοινωνικά στρώματα είναι σημαντικό να, να προσεχθούν. Επίσης, η τυπική και η άτυπη εκπαίδευση θα πρέπει ειδικά να προωθηθούν. Στα κράτη-μέλη υπάρχουν διαφορές μεταξύ, πολλές φορές μεταξύ Υπουργείου Παιδείας και Υπουργείου Πολιτισμού γιατί η προβληματική των νέων δεν μπορεί να ενταχθεί μόνο ε, στα πλαίσια κάτω από την πολιτική της ε, εκπαίδευσης, ε, της παιδείας. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρχουν ειδικά προγράμματα για νέους. Ίσως ε, λοιπόν θα μπορούσε το υπάρχον πρόγραμμα να γίνει ένα υποπρόγραμμα ε, στα πλαίσια αυτά να γίνει για τους νέους. Ευχαριστώ. Θα πρέπει να φύγει ε, σύντομα η Επίτροπος, οπότε μη μακρηγορείτε. Ε, θα συζητήσουμε εκτενέστατα το θέμα του χρόνου. Μη στενοχωριέστε. Ένα λεπτό θα δίνω στον καθένα. Η κυρία Παλιαδέλη. Ναι, ε, yes, yes, I will. Ε, ευχαριστώ να συμπληρώσω και εγώ για τα θετικά στοιχεία αυτής της πρότασης, κυρία Επίτροπε. δύο σύντομες ερωτήσεις. Ε, δεν βλέπω πουθενά την, την έρευνα σε σχέση με την εκπαίδευση Βεβαίω η έρευνα είναι ένα άλλο κομμάτι, αλλά έχω την αίσθηση ότι πρέπει να περιληφθεί και η έρευνα μέσα στην ε, εκπαίδευση, γιατί τα πανεπιστήμια κάνουν και τα δύο πράγματα. Επίσης δεν βλέπω και ελπίζω να ε, περιληφθεί ε, η πολιτιστική κληρονομιά, cultural heritage, μέσα στο culture. Γιατί βλέπω πολύ μεγάλο ποσό για, το, για τα media, για παράδειγμα, και μειωμένο το ποσό για το culture, στο οποίο φαντάζομαι ότι περιλαμβάνεται το cultural heritage. Έχω την αίσθηση δηλαδή... Ε, δεν ξέρω, συγγνώμη, έκανα λάθος, αφήστε το αυτό. Ναι. Λοιπόν, ε, πιστεύω επίσης ότι πρέπει να υποστηρίξετε τις υποδομές στα πανεπιστήμια. Δεν ξέρω με τι πρόγραμμα, είναι ένας από τους τρόπους που θα επιτρέψουν την ε, αναβάθμιση και ελπίζω ότι μέσα σε αυτό θα είναι και οι ανθρωπιστικές σπουδές και η υποστήριξή τους και στο ερευνητικό και στο διδακτικό επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Äh, Ευχαριστώ, κυρία Τρίπελ. Ευχαριστώ. Φαίνεται ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι περίθυμο. ε, φιλο, φιλότιμο και είναι, έχει μεγάλες προοπτικές, αλλά εάν δεν υπάρχουν χρήματα για αυτό το προϋπολογισμό, δεν θα πρέπει να μπορέσουμε τίποτα να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Πώς θα κάνουμε πραγματικά τις πληρωμές εφόσον υπάρχουν δεσμεύσεις. Θα πρέπει να το δούμε αυτό το πράγμα, γιατί βρισκόμαστε ενώπιον δίσκων ε, κατάσταση ενώπιον η οποία βρισκόμαστε λόγω της παρούσης κρίσης. Είπατε είπατε μία οργάνωση για κάθε χώρα. Και είπατε από επιχορηγήσει σε δάνεια. Τι αυτό σημαίνει, κύριε Κώστα παρακαλώ. Πάρα πολύ σύντομα πρόεδρε. Φυσικά, είπατε, καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά και υποδέχομαι αυτό το στρατηγικό σήμα το οποίο δίνεται όσον αφορά τι, το είπε πάρα πολύ καλά ο Επίτρο, Επίτροπος πολύ καλά και το είμαι πολύ αποφασιστικότητα διότι αυτό το education, το εκπαιδευτικό, θα πρέπει να δούμε κα, πώς θα βρούμε σε αυτό το ε, ένα τρόπο να καλύπτει όλους τους τομείς και αυτό θα μπορούσε να ε, πάρει ένα άλλο όνομα και να γίνεται Σοφία για παράδειγμα που είναι η Σοφία. Έτσι λοιπόν θα πρέπει, ελέγχθηκε προηγουμένως και πρέπει να πούμε θα πρέπει να υπάρχει το όνομα Εράσμος το οποίο είναι ένα σήμα κατά τεθένα. Υπάρχουν και τα Λεωνάτο, υπάρχουν και άλλα προγράμματα. Ωστόσο θα πρέπει, δεν πρέπει να δούμε όχι ποια, ποια τα διοικούν, ποια τα διακυβερνούν, αλλά αυτοί οι οποίοι πραγματικά εκμεταλλεύονται, δίνουν, έχουν τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν. Θα πρέπει να υπάρχει ένας τέτοιος προσανατολισμός τέτοιο, σε αυτούς όλους, ότι δεν νομίζω αυτή τη στιγμή απλοποιήθηκαν τα σχέσει εντό τη ε, ΕΕ. Είναι απλοποίηση για αυτούς που είναι από πάνω, θέλετε, και για αυτούς οι οποίοι θα κάνουν το αίτημα. Αυτή είναι μια άποψη την οποία έχω εγώ. Εγώ θα ήθελα να μην εξαφανιστεί η λέξη ε, κρεατιβιτά, δημιουργία σε σχέση με την λέξη κουλτούρα που είναι ή πολιτισμό. Η, η λέξη κουλτούρα είναι πολύ πιο μεγάλη από τη λέξη δημιουργικότητα και εγώ ανησυχώ για αυτό το πράγμα ότι αυτά τα δύο. Ποιο είναι το απτό αυτό ε, σημείο το οποίο ε, μπορεί να γραφεί εδώ μέσα. Το οποίο είναι αυτό και όχι να είναι θεωρητικό. Ευχαριστώ. Επόμενη. Ευχαριστώ. πολύ και θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Επίτροπο. Νομίζω ότι κάνατε καταπληκτική δουλειά. Έχω κάποια σχόλια για το πρόβλημα με τις ονομασίες, γιατί βλέπω ότι αυτό όλους μας ε, ανησυχεί. Είναι και κάπως ανόητο όταν έχουμε τόσο γνωστά εμπορικά σήματα να μην τα χρησιμοποιούμε. Φαντάζομαι λοιπόν πως όταν θα ξεκινήσουν όλα αυτά τα προγράμματα υπό το ενιαίο πρόγραμμα θα έχετε γραμμές ε, για το καθένα στον προϋπολογισμό. Άρα θα εξακολουθήσει να υπάρχει γραμμή πούμε για το Marie Curie, για το Comenius. Δηλαδή θα έχετε κάποιο τρόπο να εξασφαλίσετε ότι υπάρχει φάκελος που θα δοθεί σε συγκεκριμένο σκέλος του προγράμματος. Γιατί λοιπόν δεν θα μπορούν να συνεχίσουν ως υποπρογράμματα και να εξηγήσουμε στους ετούντες ε, ότι συμβαίνει αυτό για να διατηρήσουμε τις ονομασίες και να τους πούμε εντάξει θα ζητήσετε χι για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ε, μια πρακτικής φύσης ε, πρόταση γιατί πραγματικά πιστεύω ότι το όνομα κάνει τη διαφορά και θα πρέπει να βρούμε ένα γενικότερο όνομα ομπρέλα κάπως διαφορετικό. Ε, πριν ληφθεί η απόφαση, σας παρακαλώ πολύ, συμβουλευτείτε μας. Γιατί αυτό το οποίο θα δώσετε ως όνομα θα επηρεάσει και τη μελλοντική του επιτυχία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο και εγώ στον εαυτό μου δεν θα, κάνουμε, δεν θα γίνουν διαβουλεύσεις με εμάς. Εμείς θα αποφασίσουμε, εμείς από κοινού θα αποφασίσουμε πώς θα ονομαστεί. Το lifelong learning ε, τώρα είναι γενικότερη έννοια. Το Erasmus for All δεν είναι γενικότερη έννοια, γιατί εστιάζει σε ένα κομμάτι, την κινητικότητα, που συνδέεται με τα πανεπιστήμια. Ε, έχει δίκιο κυρία Κάμεραϊν, τα δημοτικά και τα γυμνάσια δεν μπορούμε να τα βάλουμε να ανταγωνίζονται την τροβάθμια εκπαίδευση. Εμείς θέλουμε ε, να ισχύουν τα ποσοστά και όντως να μεταφραστούν ε, σε περισσότερα χρήματα, αλλά τα, νούμερα που έχω εγώ ε, δείχνουν ότι το minimal allocation, η ελάχιστη δηλαδή προοικοδότηση, αν πάρουμε ας πούμε τριτοβάθμια, είναι 58% του συνολικού προγράμματος. Πού είναι, πού πάνε τα υπόλοιπα 40, το υπόλοιπο 42%. Δεν ε, επιτρέπω σε κανέναν να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες χωρίς να διαβουλεύεται με το Κοινοβούλιο. Και αν ε, συνεχίσουμε έτσι, δεν θα μας ρωτήσει κανείς τι θα γίνουν τα υπόλοιπα χρήματα, γιατί θα υπάρξει επιτροπολογία μεταξύ Συμβουλίου και Επιτροπής. Και αυτό δεν επιτρέπεται. Σταματώ, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Επίσης, στο πρόγραμμα, πού είναι η Μπρουζ, πού είναι η Φλωρεντία, ε, για παράδειγμα. Αυτά πρέπει να τα ξέρουμε. Είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε ιδρύσει το Ζαν Μονέ το βρήκα. Και κάτι ακόμα. Δεν ξέρω με ποιους ε, εμπλεκομένους ε, μίλησε η Κομισιόν. Όλοι οι εμπλεκόμενοι που ήρθαν στο γραφείο μου και που του συνάντησα αλλού ε, έλεγαν ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει το γενικό έμβλημα Εράσμους. Το lifelong learning είναι η γενική έννοια που μπορεί να τα εντάξει όλα. Ε, μπορούμε να το διαπραγματευτούμε αυτό. Εάν δημιουργήσουμε ένα καινούριο ε, όνομα, ε, αυτό θα πρέπει να το συνεννοηθούμε. Επίσης, για την, τα loans και grants για τις δημιουργικές τέχνες, ήμουν στο Μόναχο στις ε, ημέρες, ημερίδες των ΜΜΕ ε, μας είπαν για τα δάνεια εντάξει, αλλά τις εγγύσει για τα δάνεια θα τις αναλαμβάνουμε εμείς και όταν θα πρέπει να ε, ενεργοποιηθούν οι εγγύσει, θα πληρώσουμε εμείς από τον προϋπολογισμό για τον πολιτισμό. Ε, οπότε ε, πολύ γρήγορα θα διάσουν τα ταμεία μας. Εδώ χρειάζεται μεγάλη προσοχή, αλλά θα χρειαστεί οπωσδήποτε να ξανασυζητήσουμε στο... του χρόνου για αυτό το θέμα. Περιορίζομαι λοιπόν εδώ και δίνω το λόγο αμέσως στην Επίτροπο. Ευχαριστώ. Καταρχήν επιτρέψτε να σας πω τα εξή. Σέβομαι τα προνόμια τα οποία έχετε να και εσείς θα αποφασίσετε βεβαίως, δεν θα ζητήσω αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή και πιστεύω ότι θα είμαι η τελευταία η οποία ότι δεν λαμβάνω υπόψη μου αυτό το κοινοβούλιο και αυτή την επιτροπή υπόψη μου. Νομίζω πως τα πράγματα θα γίνονται πάρα πολύ δημοκρατικά και νομίζω πως εδώ υπάρχει δημοκρατία και σε αυτή την επιτροπή. Επιτρέψτε μου τώρα να σας πω από την αρχή ότι υπάρχει μια παρεξήγηση όσον αφορά το Marie Curie. Αυτό δεν βρίσκεται, Μαρικύρη δεν βρίσκεται μέσα σε αυτή την ομπρέλα. Είναι στον ορίζον το 2020 και υιοθετήθηκε την επόμενη και παλεύω για να πάρω περισσότερα χρήματα για το Marie Curie και νομίζω πως πραγματικά θα προσπαθήσει, πρέπει να προσπαθείτε και να με υποστηρίξετε. Και υπάρχει μια πρόταση για να τροποποιήσουμε όλα αυτά με με, βλέποντας πραγματικά από πού έρχεται η Μαρικυρία όταν είναι Πολωνή στην καταγωγή. Τώρα, όσον αφορά την απλοποίηση, ας είμαστε σαφείς από την αρχή, εγώ ζήτησα αυτό το πράγμα. Εάν θέλω πραγματικά να έχω περισσότερα χρήματα, θα πρέπει να το ίσου να γίνει αυτή η τεμαχιοποίηση του προγράμματος. Και βεβαίως οι επιλογές μου ήταν πολύ περιορισμένες αντί να αποφασίσω για το Erasmus φορολό, All, ε, αποφάσισα ένα άλλο πρόγραμμα, αλλά θα πρέπει να καταργήσω όλα Κρούντφιχε, Λεωνάρντο, Youth in Action, όλα αυτά τα προγράμματα θα πρέπει Εράσμους Πουρτούς νομίζω ε, Βάζω τα διεθνή του ονόματα που είναι αγγλικά, γαλλικά και το καθεξή για να απλοποιήσω, λέει ο Μήτριο. Η επιλογή μου λοιπόν ήταν περιορισμένη. Επέλεξα λοιπόν εκείνο το όνομα που κατά την ακρίση μου μπορεί να έχει διαφορετική εντύπωση όταν ταξιδεύω οπουδήποτε εντός της ε ή εκτός έχει ένα όνομα το οποίο έχει στο στόμα του καθενός. Ακόμη και οι συνάδελφοί μου να παίρνουν το όνομα Εράσμου στη συνάδελφοί μου της Κομισιόν για άλλο λόγο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ποιε ήταν οι επιλογέ, ποιες ήταν οι επιλογές που πρέπει να κάνουμε. Το ελάχιστο της, ε, της παροχής αυτή τη στιγμή είναι για να προστατεύσουμε τους διάφορους τομείς. Ανησυχείτε βέβαια εσείς για τους νέους. Ε, εγώ βεβαίω ανησυχώ ακόμη περισσότερο διότι όλα τα προγράμματα αυτά έχουν εστιάζονται επί των νέων. Επίσημη, ανεπίσημη εκπαίδευση. Και αυτό στους διάφορους τομείς είπα εγώ και επανέλαβα ότι δεν θέλουμε μία νέο οργάνωση ε, οργάνωση φοιτητική, οποία, η οποία θα είναι μεγάλη μικρή και η οποία θα ανταγωνίζεται με το πανεπιστήμιο. Έτσι λοιπόν αυτό είπαμε που θα γίνει είναι για διάφορες κατηγορίες θα υπάρχουν παροχές οι οποίες υψηλή, ανωτέρη εκπαίδευση, κατάρτιση, επαγγελματική κατάρτιση, έχουμε τους νέους, έχουμε άλλες υποκατηγορίες και έχουμε την διεθνή διάσταση. Όλα αυτά, εάν τα δείτε και δείτε ποια είναι το ελάχιστο ε, ε, των χρημάτων που γίνεται, είναι ένα ποσό το οποίο είναι από τα που θα πάρουμε από το προπολογισμό που έχουμε σχεδιάσει. Αλλά δίνει τη δυνατότητα ακόμη να, να αποφασίσουμε μαζί κάθε χρόνο ποια είναι η δυνατότητα απορρόφησης από όλους αυτούς τους αναφερθέντες τομείς και να κάνουμε τις παλαιοφ... Πόσο θα πάει εκεί, σύμφωνα με την ζήτηση που θα υπάρξει. Το ετήσιο πρόγραμμα θα συνεχιστεί λοιπόν θα προταθεί και θα συμφωνηθεί ομού μεταξύ μας, σύμφωνα με τις, με τις αιτήσει και τις προτεραιότητες που θα υπάρξουν. Ο κ. Λόκερχαντ αναφέρθηκε στι εξωτερικέ σχέσει μας και αυτή την ισορροπία η οποία υπάρχει μεταξύ των ανταλλαγών φοιτητών, μεταξύ ε, Ευρώπης και Κίνας. Πριν δεν μου ήμουν εγώ στην Κίνα και συμφώνησε με την κοινωνική κυβέρνηση ότι έχουμε διορίσει τους πιο υψηλό ε, επίπεδο. Είναι μια κυρία η οποία βρίσκεται στο πόλο του Πουρό της Κίνα και ε, βεβαίω ο τρίτος πυρώνας ε, των σχέσεων όταν ο πρόεδρος της Κίνας και του Μπαρόζο θα είναι ήταν εκεί αλλά αναβλήθηκε άλλα, νεολαία, εκπαίδευση κλπ. Πολιτισμό, όλα αυτά περιλαμβάνουν στον τρίτο πυλώνα των σχέσεων με την Κίνα. Και σε αυτό το σημείο προκύπτει για το Εράντους Μούντους και Τέμπους και όλα αυτά τα άλλα προγράμματα, όλα αυτά συμπεριλαμβάνουν σε ένα και δίνουν, δίνουν τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή στους νέους μας να κάνουν αίτηση για το Εράσμος και να πάνε σε ένα άλλο πανεπιστήμιο, στην Κίνα, στην Ιαπωνία ή στη ΣΥΠΑ. Ανοίγουμε λοιπόν και για τις γειτονικέ μας χώρες ακόμη. Και βέβαια θα υπάρχουν και άλλα προγράμματα, κοινά προγράμματα για PhD, για masters, για δοκτορά δηλαδή. Υπάρχουν λοιπόν τεράστιες προοπτικές σε αυτό το τομέα. Τώρα κάτι άλλο. Πολλά μέλη εξέφρασαν την ανησυχία τους όσον αφορά δομικές, τα δομικά γεγονότα. Αρκεύει πως πραγματικά η κουλτούρα και το σπορ δεν αναφέρονται. Ε, ωστόσο, έχουν στα διαθετικά τα, ε, ταμεία τη δυνατότητα αυτή διότι σκοπός όλων αυτών των ταμείων είναι μέχρι το 20 να εξυπηρετήσει αυτού τους στόχους. Διότι το σπορ είτε χρειάζεται ένα στάδιο, είτε ένα πανεπιστήμιο να κτιστεί, είτε να εξυγχρονιστεί ή ένα, μια εκδήλωση καλλιτεχνική να γίνει, όλα αυτά τα πάρουμε από τα διευθυντικά ταμεία και όλα αυτά στην πολιτική και στη στρατηγική μέχρι το 2020. Κάτι άλλο. Το, η πολιτιστική κληρονομιά βεβαίω είναι ένα μέρος του, του πολιτισμικού μας προγράμματος. Μην ξεχνάτε αυτό που γίνεται κάθε χρόνο και αυτό θα συνεχιστεί για την κληρονομιά οι μεταφράσεις των φιλολογικών κειμένων, τα πολιτισμικές εκδηλώσεις θα συνεχίσουν να υπάρξουν και ακόμη σήμερα γίνονται και θα γίνονται κάτω από το κεφάλαιο πολιτισμικών εκδηλώσεων που γίνονται εκ μέρους μας. Βεβαίως έχουμε περισσότερα χρήματα για τα μίντια από ό,τι για την κουλτούρα, γιατί τα μίντια κοστίζουν πολύ περισσότερο. Έτσι δεν είναι. Έχουμε επίσης μία νέα φάση, μία νέα, ένα στρώμα και αυτό θα, διε, θα βοηθήσει περισσότερο για δάνεια πολιτισμικά τα οποία δίνονται και, και σε αυτό το σημείο είπα ότι πραγματικά χρειαζόμαστε, ναι, ναι, Εκεί είπα ότι πρέπει από επιχορηγήσεις θα πάμε σε loans, σε, σε δάνεια θα υπάρχει, θα υπάρχει εγγύηση για τα δάνεια τα οποία, τα loans. Αλλά η μόχλευση αυτή θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Το κέρδος που θα προκύπτει θα είναι πολύ μεγαλύτερο. Εάν όχι, φοβάμαι ότι πρέπει να φύγω γιατί έχω μια ε, συνδιάσκεψη τύπου, διάσκεψη τύπου αλλά νομίζω πως πραγματικά θα έχουμε ξανά την ευκαιρία να ξανασυζητήσουμε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και πρέπει να φύγω. Γεια σας, ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι έχουμε πολλές, θα έχουμε πολλές συζητήσεις, ήδη από το Γενάρη θα έχουμε και θα αποφασίσουμε ποιος θα είναι εισηγητής γιατί. Βεβαίως έχουμε διαφορετικές απόψεις εδώ μεταξύ μας και θα τα συζητήσουμε. Εγώ, πολύ, εγώ περισσότερο με αγγίζουν, για μένα με τα πράγματα εκείνα τα οποία πρέπει να αλλάξουν και, και βεβαίως χαίρομαι πάρα πολύ για τους στόχους οποίους έχονται. Έτσι περαιτέρνουμε. Όχι. Γεια σας, κύριε Επίτροπε. 12 σημείο θα πρέπει Είναι κατά κανεί των, των συντονιστών χθες. Όχι. Υπάρχει τίποτα άλλο. Θέλει κανείς any, any business να πάει στα διάφορα. 20-21 Δεκεμβρίου είναι η τελευταία μα συνεδρίαση πριν από τα Χριστούγεννα. Είναι κανείς εναντίον? Όχι. Λαμπρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πέρα συνεδρίαση.